Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose de commencer. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Και προτείνω να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε, συζητώντας το θέμα 1, την έγκριση δηλαδή, ε, θα σας πρότεινα λοιπόν να δούμε αυτή την πρόταση του Συμβουλίου για τον κανονισμό το σχετικό με, τον, με την αντικατάσταση του 843 του 2004 και του 2049 του 2009 ε, για τους υπηκόους κρατών που δεν καλύπτονται ακριβώς λόγω διαφορετικής ηθαγένειας από τους κανονισμούς και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εξέταση της κοινής θέσης του Συμβουλίου στα θέματα αυτά που θα πρέπει να συζητηθούν στη συνεδρίασή μας. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση. Θα προσθέτουμε λοιπόν στην ημέρηση διάταξη στα πρακτικά της συνεδριάσεως της 23-24 Ιουνίου. Πάλι δεν βλέπω παρατηρήσεις. Άρα θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν. Ανακοινώσει. Καταρχά ανακοινώνω ότι ελπίζω να έχετε περάσει καλέ διακοπές. Και δεύτερον, πιο σοβαρά, με χαρά καλωσορίζουμε μεταξύ μας νέο μέλος της Επιτροπής μας, τον κύριο Σέρτζο Γκουτιέρε Πριέτο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες που αντικαθιστά ως αναπληρωτής τον κύριο Περέιο, ο οποίος δεν είναι εδώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι εδώ, ε, του ευχόμαστε εξ αποστάσεως και τηλεπαθητικά το καλώς όρισες. Όσοι ήθεστε, ήθιστε έχουμε μετάδοση ε, μέσω του ίντερνετ της συνεδριάσεως. Άρα μπορεί να μας παρακολουθούν και από το ίντερνετ και θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμα η ανακοίνωση σχετική με την αποστολή της ε, Επιτροπής μας στο Δουβλίνο και το Λίμερικ 2 και 4 Ιουνίου ανακοίνωση την οποία έχει ετοιμάσει η Γραμματεία, θα δείτε στους φακέλους σας και υπάρχει θέση σας στις ε, τρεις γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά. Ακόμη δύο ανακοινώσεις στο ίδιο πνεύμα. Η μία έχει να κάνει με την ε, εκδήλωση στο Παλέντεγμό στις Βρυξέλλες για την προετοιμασία της Βελγικής Προεδρίας και δεύτερη ανακοίνωση η σχετική με την άτυπη συνεδρίαση της ΕΠΣΚΟ τον Ιούνιο, όπου εκπροσώπησα εγώ την Επιτροπή μας, ιδίως σε θέματα συζήτησης ε, κυρίως, ε, σε θέματα που συζητήθηκαν κυρίως με τον ε, Πρόεδρο κύριο Φαν Ρόμποϊ. Επίση, η συζήτηση που έπρεπε να γίνει μέσα στην Επιτροπή μας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μελετών ε, αντικτύπου ως προς την άδεια μητρότητας και τις κινητοποιήσεις σχετικές με τις απεργιακές ε. όχι λοιπόν, ξαναρχίζω. Τις ε, απεργίες κατά της μεταρρύθμισης στη Γαλλία του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων μας υποχρέωσαν αυτές οι απεργίες να αναβάλουμε για μεταγενέστερη ε, ημερομηνία αυτή την συνάντηση και το εργαστήριο για την αδιαπληκτρότητα προς το θέλει του μήνα δηλαδή θα σας ενημερώσω και επίση πρέπει να σας ενημερώσω ότι η έκθεση ορί πρόκειται να ψηφιστεί, ε, πρόκειται να ψηφιστεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια Εγώ ε, φρόντισα να έρθω σε επαφή με την ε, κυρία Μιλικέ, η οποία είναι η πρόεδρος ε, της ομάδας ΕΠΣΚΟ, για να της εξηγήσω, τις, η προεδρεύουσα της ομάδας ΕΠΣΚΟ, για να της εξηγήσω τις θέσεις μας πριν από τις θερινές διακοπές ακόμη, να πω ποιε είναι ακριβώς οι προτιμήσεις και τα σημεία στα οποία αντιδρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ληφθούν αυτά υπόψη κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου, δεδομένου ότι η ομάδα εργασίας, ΕΠΣΚΟ, πρόκειται να συνεδριάσει αύριο. Η γραμματεία της κυρίας Μιλκέ με ενημέρωσε ότι όντως έλαβε τη σχετική επιστολή μου και ενημερώνει ε, τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στο Συμβούλιο για τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ελπίδα μια παραγωγική και αποτελεσματική ε, κατάληξη να προκύψει βάση των θέσεων του Κοινοβουλίου. Μάλλον έχω ολοκληρώσει τις ανακοινώσεις μου τώρα. Και ως εκ μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Καταρχάς καταγράφουμε, λαμβάνουμε γνώση της κοινής θέσεως που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο για τον κανονισμό 997-2009 για τους ε, υφικούς τρίτων κρατών που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές μόνο και μόνο λόγω ηθαγενείας. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ ήταν η ε, αρμόδια για την έκθεση αυτή όταν ε, την είχαμε. Δεν ξέρω αν θα πείτε κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να κάνω και εγώ μία ανακοίνωση στην Επιτροπή αυτή και να συνημερώσω για την απάντηση προς το Συμβούλιο. Υπάρχει μία καταλεκτική ημερομηνία που έχει δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για, την, για τον ίδιο τον κανονισμό αυτή τη στιγμή. Να κάνω και μια, κάποιες προτάσεις και οι συνάδελφοι μπορούν να σκεφτούν περισσότερο τις προτάσεις αυτές στη συνέχεια. Ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κανονισμός που έχει να κάνει με την διασυνοριακή κατάσταση όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση για επικόους τρίτων χωρών που πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη, από ένα κράτος μέλο στο άλλο. Στόχος λοιπόν του νέου σχεδίου κανονισμού είναι να επικαιροποιήσει την κατάσταση, καθότι έχουμε προχωρήσει σε, στην εφαρμογή ενό κανονισμού όσον αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση ήδη από πέρυσι. Στην πρώτη λοιπόν ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Προσπαθήσαμε να δούμε πώς είναι η νομική βάση, η οποία τώρα έχει τροποποιηθεί. Επομένως, η πρόταση διαβούλευση που είχαμε κάνει πέρασε ως τοποθέτηση πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάνουμε ουσιαστικά δύο προτάσεις τροποποιητικές ως προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να επανέλθουν πάλι δύο ρήτρε οι οποίες αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης. Το Συμβούλιο δέχτηκε τις δύο αυτές προτάσεις, τις δύο αυτές τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι ε, Θα υπάρχουν πολλές τροπολογίε από πλευρά του Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την νομική βάση άρθρο 79β. Η Δανία δεν συμμετέχει καθόλου στο νέο προβλεπόμενο καθεστώ, όσον αφορά τους υπηκόου τρίτων χωρών που κινούνται διανοστεριακά από τη μία χώρα στην άλλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Δανία έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει καθόλου στο πακέτο αυτό μέτρων που αφορούν του ε, υπηκόου τρίτων χωρών. Δυστυχώ επίση και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην επικαιροποιημένη, ε, στον επικαιροποιημένο κανονισμό. Θα ισχύει λοιπόν ο παλαιότερο κανονισμό για αυτού και η Ιρλανδία αποφάσισε επίση ότι δεν θα συμμετέχει. Επομένως, πολλές τροπολογίες που υπάρχουν ήδη στην τοποθέτηση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζουν την κατάσταση αυτή ως έχει. Ότι υπάρχουν δηλαδή κάποιες χώρες οι οποίες ε, επιθυμούν να μη συμμετέχουν, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, και βέβαια το καθεστώς αυτό δεν βοηθάει καθόλου την απλοποίηση του κανονισμού όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση των υπηκών τρίτων χωρών που κινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, που κινούνται διασυνοριακά. Πολύ σύντομα θα υπάρχει ένα έγγραφο επίσημο με τις συστάσεις μου, όπου θα λέγεται ότι μπορούμε να δεχθούμε το κείμενο του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο από την Βελγική Προεδρία, ενδεχομένω στα πλαίσια τη Τρόικα, ένα εκπρόσωπο τη Ισπανική Προεδρία θα μπορούσε να πει κάτι όσον αφορά την επίτευξη συμφωνία στο Συμβούλιο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι το να φτάσουμε σε μια κοινή θέση δεν ήταν και τόσο εύκολο χρειάστηκε να αλλάξει η νομική βάση της συνθήκης και να περάσουμε από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Δύο φορές το Συμβούλιο προσπάθησε να εγκρίνει το κείμενο αυτό και τις δύο φορές δυστυχώς λόγω της αντίρρησης κάποιων χωρών δεν εγκρίθηκε. Περνώντας λοιπόν στην ειδική πλειοψηφία επιτρέψαμε να υπάρχει μία οδός που ακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια του περασμένου εξαμήνου. Δηλαδή η ιδέα μας ήταν να εγκρίνουμε έναν κανονισμό συνενετικό αρχικά με το Κοινοβουλίο και αυτό ακριβώς κάναμε. Πάντοτε πριν από τις συναντήσεις με το Συμβούλιο δηλαδή συζητήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια σύγκληση. Δεύτερον, η βασική ιδέα ήταν ότι στους υπηκόους τρίτων χωρών θα έπρεπε να εφαρμόσουμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις και χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τις παροχές. Και τρίτον, ουσιώδες κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να αφαιρέσουμε τις εξαιρέσεις που περιλάμβανε ο κανονισμός 859. Γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους θα δείτε ότι εγκρίναμε ένα κείμενο με την θέση τριών χωρών και την αποχή μιας άλλης χώρας που είναι πολύ σύντομο είναι ένα κείμενο το οποίο το μόνο που λέει είναι ότι ο νέος κανονισμός 883 θα εφαρμόζεται και για τους υπηκόους των τρίτων χωρών. Και μιας και έχω το λόγο, να σας παρακαλέσω κάτι. Από την 1η Μαΐου 2010 εφαρμόζεται ο κανονισμός 883. Όταν παλαιότερα είχαμε εφαρμογή αυτού του κειμένου μπορούσαμε να εφαρμόζουμε και τον κανονισμό αυτό για τους υπηκόους των τρίτων χωρών. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό διαφορετικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών θα εφαρμόσουμε ένα νομικό εργαλείο διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζουμε για τους κοινοτικού υπηκόους. Γι' αυτό ακριβώς ζητώ μια έγκριση ταχεία, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να ενοποιήσουμε το κείμενο και από την έγκριση του κειμένου αυτού να εφαρμόσουμε το 883 κανονισμό και στους κοινοτικού αλλά και στους υπηκόους των τρίτων χωρών. Τέλος, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λαμπέρτ, περιλάβαμε τις τροπολογίες που είχε καταθέσει το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό αρχικά και σε σχέση με την μη εφαρμογή εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου του νέου κανονισμού νομίζω και αυτό βεβαίω είναι μια εκτίμηση καθαρά προσωπική ότι τελικά έστω και να έχουμε να κάνουμε με επίπεδο διοικητικών διαδικασιών θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μια χώρα να εφαρμόσει ένα κανονισμό και οι υπόλοιπε χώρε να εφαρμόσουν ένα άλλο. Όπω έλεγα προηγουμένω, σε επίπεδο διοικητικών διαδικασιών, μελλοντικά προβλέπω μια σύγκληση μεταξύ τη εφαρμογή που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και τη εφαρμογή που κάνουν όλε οι υπόλοιπε χώρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο πρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στην ανακοίνωση που εστάλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την συμβαστική λύση που βρέθηκε στο Συμβούλιο. Η κοινή θέση συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που υπήρχαν αρχικά και στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει επίσης τις δύο τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν σε πρώτη ανάγνωση και περιλαμβάνει τι τροποποιήσει εκείνε που έχουν ω στόχο να διευκρινίσουν, να απλοποιήσουν κάποιε ρήτρε, κάποιε διατάξει. Και όπω υπόθηκε, ο νέο κανονισμό ε, συντονισμού ισχύει για του ε, υπηκόου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι αυτοί οι όροι να μπορούν να ισχύουν και του υπηκόου τρίτων χωρών. Λέει ο σύντομα να πω ότι είναι σωστό να πούμε ότι θα πρέπει να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο την Ισπανική Προεδρία αλλά και τη Βελική Προεδρία ώστε να προχωρήσει αυτός ο φάκελος και να είναι εφαρμόσιμος και να εφαρμοστεί και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που πραγματικά αντιμετωπίζουν μια κατάσταση διακρίσεων να πω κατά δεύτερο λόγο ως κοιόδης εισηγητής από την σοσιαλιστική ομάδα και να πω στην σύντροφο Λάμπερτ ότι είμαστε σε θέση επειδή ακριβώς οι κυριότερες θέσεις του Κοινοβουλίου έγιναν δεχτές από την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο να πω ότι όταν θα είναι έτοιμη η έκθεση εμείς θα την δεχτούμε θετικά και γι' αυτό ακριβώς συμφωνούμε με το αίτημα που υποβλήθηκε προηγουμένως να τελειώνουμε όσο γίνεται νωρίτερα με το θέμα αυτό, επειδή ακριβώ υπάρχει αυτό το νομικό κοινό το οποίο ισχύει από την 1η Μάη του 2010. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Λάμπερτ, θέλετε να λάβετε και πάλι το λόγο. Όχι, κύριε Όμεν. Ναι, Πρόεδρε. Εγώ ήμουν η συντάκτης της τροπολογίας και θα ήθελα ξεκάθαρα να αναφέρεται στην νέα νομοθεσία ότι δεν υπάρχουν ε, παρεκκλήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη αυτό να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις δηλαδή ως προς την απαγόρευση ε, των γενετικά τροποποιημένων αυτών οργανισμών. Και άπαξ και υπάρχει αυτό, βρίσκουμε λύση για τα πάντα. Très bien, Madame Lambert. Κύριε Λέμπερτ, Για να απαντήσω στην παρατηρήση της κυρίας Σόμεν, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν προβλέπονται παραρτήματα έξω, όσον γνωρίζω. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, από ό,τι φαίνεται, έχει συμπεριληφθεί ως είχε, άλλωστε το Κοινοβούλιο δεν είχε ψηφίσει καμία εξαίρεση, αυτή είναι θέση μας. Και από ό,τι ξέρω, το ψήφισμα ενσωματώνεται στην νομοθεσία. Αυτό γνωρίζω εγώ. Βέβαια θα το επιβεβαιώσω πριν την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή και σε συνεργασία με τους πιο δυσηγητές. Ε, ε, Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Θα περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Καταρχάς, θα ψηφίσουμε για το σημείο 4, θέση του Κοινοβουλίου η δική μας τουλάχιστον συνεισφορά όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού για το 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο όλα τα τμήματα. Σημείο 4 λοιπόν, όπως σας είπα, θα ψηφίσουμε για την ε, θέση μας όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού για το 2011, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε αρχικά τις ε, τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τα ποσά 0401-01 Μία πρώτη τροπολογία. 6.301 κυρίας Μπάστος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Έχετε όλη την κάρτα σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχετε, έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ψηφίσατε πέρας. Προσπαθήσατε να βγάλετε και να ξαναβάλετε την κάρτα σας. Προτείνω να ψηφίσετε σηκώντας το χέρι σας, αλλά από ό,τι βλέπω λειτουργεί, λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 21 κατά, δεν εγκρίνεται, απορρίπτεται. Τροπολογία 6300 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ατροπολογία. 63-33 υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Le vote est... Πέρας. 15 υπέρ. 21. Κατά. Απορρίπτεται. Επόμενη γραμμή, τροπολογία 6.302 της κυρίας Μπάστος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6.334, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλω να σας πω απλώς ότι ε, κατά αυτόν τον τρόπο δεν ψηφίσαμε καμία τροπολογία για να επανέλθουν κάποιες γραμμές στο νέο προπολογισμό και αποδεχόμαστε αστικά όλες τις περικοπές του, που προτείνει το Συμβούλιο. Το ΕΛΚ δεν κατάφερε να πετύχει να περάσει την δική του αύξηση, αλλά ούτε και εμείς αυτή τη στιγμή. Επομένως τα πράγματα παραμένουν ακριβώς όπως το πρότεινε το Συμβούλιο, μολονότι ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες υπήρχε αν μη τι άλλο μια πλειοψηφία για την αύξηση των ε, ποσών που είχε αρχικά προτείνει το Συμβούλιο. Εμείς τώρα με την ψηφοφορία που κάνουμε δίνουμε στο Συμβούλιο το δικαίωμα να διατηρήσει το κείμενό του και να μην γίνει καμία αύξηση. Σας το λέω αυτό απλώς αυτή τη στιγμή, να το έχετε κατά νου. 6.335 η τροπολογία η οποία ουσιαστικά έχει ως στόχο να επανέλθει η αρχική πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκρίνεται. 6.336 για τον ίδιο λόγο πάλι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6303 της κυρίας Μπάστος. Μάλλον να κάνουμε πρώτα ηλεκτρονικό έλεγχο για το 6336. Άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ. 21 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 6.303 της κυρίας Μπάστος υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 18 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 6.304 της κυρίας Μπάστος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ...6.337. Πάλι εδώ πέρα, μάλλον καταπίπτει, με συγχωρείτε, γιατί εγκρίναμε την 6.304. Περνάμε στην τροπολογία 6338 για να επανέλθουν οι αρχικές γραμμές του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.305 της κυρίας Φιγκερέντο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6.307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6.306 της κυρίας Μπάστος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 6.339 και περνάμε στην 6.308 υπέρ εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως και για το σχόλιο που ακολουθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 6.340 και περνάμε στην 6.309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχόλιο που ακολουθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Nous en venons Πληροφόρηση προς τους εργαζόμενους 6.311 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6.310, η τροπολογία αυτή είναι δικιά μου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.312 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 6.312. άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε και το σχόλιο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 6.342 καταπίπτει και περνάμε στην 6.313 της κυρίας Μπάστος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι ακόλουθες καταπίπτουν. Περνάμε στην 6.344 που επαναφέρει τις αρχές γραμμές επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.345 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 6.315 για ένα πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά τα μέτρα για τη διατήρηση απασχόλησης υπέρ. Οι συντονιστές είχαν συμφωνήσει γι' αυτό υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 22 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6316. Πάλι πρόκειται για συμφωνία των συντονιστών. Πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζουν οι συντονιστές για να περιέλθει στον προπολογισμό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με τις ίδιες ψήφους. Τροπολογία 6317 πάλι για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που στηρίζουν οι συντονιστές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 6.318 όσον αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα Your First Eures Job υπέρ κατά, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε και το σχόλιο το σχετικό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στροπολογία 6.320 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6.319 της κυρίας Μπάστος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας προτείνω να ψηφίσουμε και το σχόλιο της τροπολογίας 6321. Ψηφίσουμε μόνο το σχόλιο της τροπολογίας 6321 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη γραμμή του προπολογισμού που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία και ψηφίζουμε τροπολογία 6322 της κυρίας Φιγκερέντο υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 6.347 της συγγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε επίσης και το σχόλιο, το σχετικό της 6.323 υπέρ κατά αποχές. Το σχόλιο λοιπόν της τροπολογίας αυτής εγκρίνεται. Περνάμε στη γραμμή που έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας, τροπολογία 6.325 της κυρίας Φιγκερέντο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6.300 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και έχουμε εδώ πέρα και ένα σχόλιο με τρία ξεχωριστά σημεία, τρία διαφορετικά εδάφια. Σας προτείνω να το ψηφίσουμε συνολικά. Ποιο είναι υπέρ του σχολείου 6324, κατά αποχές εγκρίνεται. Γραμμή του προπολογισμού όσον αφορά το Progress. Έχουμε την τροπολογία 6326 κυρία Φιγκερέντο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6327 της συγγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχετικό σχόλιο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ισότατο των φίλων, τροπολογία της κυρία Φιγκερέντο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υποστήριξη για την εφαρμογή, τροπολογία της ηγήτριας 6.349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Εργασίας, τροπολογία 6350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Εργασία 6351 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμπλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων, τροπολογία 6352 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. πιλωτικό πρόγραμμα για καλύτερα δικαιώματα για τις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία για το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της ενδίας και του κοινωνικού αποκλεισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία για ένα πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά τον αυτισμό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι χιλιάδες της κυρίας Ήρσα πιλωτικό πρόγραμμα τους που καταλείπουν νωρίς στο σχολείο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και δεν θα ψηφίσουμε επομένω και το σχόλιο το σχετικό με την τροπολογία αυτή. Euh, Περνάμε στη γραμμή του προπολογισμού που έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια των μεγάλων εργαζομένων, δικαιωμένων εργαζομένων. Τροπολογία 6.332 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σχετικό σχόλιο με την τροπολογία αυτή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην επόμενη γραμμή. Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Τροπολογία 6357 τη ηγέτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6354 ανθρώπινη πόρη υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 6.355 Επαγγελματική κατάρτιση Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Επιδοτήσεις στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έτσι, εξαντλήσαμε τα ποσά και τα σχόλια. Μένει να ψηφίσουμε το σχέδιο χρονομοδοτήσεως. Παράγραφος 1. Τροπολογία παριθμών 3 της ηγετρίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την πρώτη παράγραφο, η υπαριθμών 4 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην του παρελθόν 5 έχει ζητήσει σε τμήματα ψηφοφορία η ομάδα του ΕΛΚΑ. Λέει η κυρία Μπερές. Θα σας εξηγήσω λοιπόν το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας, το οποίο σημαίνει ότι εισάγεται ένα βήμα υποτίθεται προς την ε, υλοποίηση αυτού του ταμείου με την πρικοδότηση με συγκεκριμένο ποσό αυτού του ταμείου, όπως άλλωστε ήταν η λογική συνέπεια των όσων ψηφίσαμε μέσα από τις γραμμές του προπολογισμού και τις εκθέσεις του κυρίου Πόρτας. Στην οποία έχει γνωμοδότηση η κυρία Μόχα. Και όπου είχε εκφραστεί ρητά το αίτημα για μια ειδική γραμμή στον προπολογισμό. Αυτά για την τροπολογία, λέει τώρα η ομιλήτρια, υπερθυμών 5. Ψηφίζουμε λοιπόν στο πρώτο τμήμα μέχρι το αγορά εργασία. Πρώτο είπε. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, τα ποσά και την γραμμή, την ιδιαίτερη γραμμή, υπέρ, κατά, αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαριθμών 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 19 κατά. Δύο αποχές. Δεν εγκρίνεται λοιπόν το δεύτερο τμήμα. Ύστερα από την τρίτη παράγραφο, τροπολογία υπαριθμών 6 της κυρίας Φιγκεϊρίδου. Προφορική τροπολογία δική μου την οποία έκανε δεκτή η συντάκτρια της τροπολογίας. Την ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, άποχες. Μάλλον έχει απορριφθεί, αλλά ας επαληθεύσουμε παρακαλώ την τροπολογία 6. Άρχιε προφορία ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 19 υπέρ 19 κατά. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 7 στην τέταρτη παράγραφο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ύστερα από την έκτη παράγραφο υπάρχει τροπολογία 10 της κυρίας Φιγκεϊρέιντο υπέρ, κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικά την τροπολογία 10 Φιγκεϊρέιντο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 9 υπέρ, 16 κατά, 11 αποχές. Δεν εγκρίνεται. Μετά την 7η παράγραφο, τροπολογία παριθμών 11 της κυρίας το υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8, τροπολογία 12 της συγκεκριτρίας υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 13 μετά την 8η παράγραφο της κυρίας το υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται. Α επαληθεύσουμε τη 13, τροπολογία 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 18 κατά. Είχατε δίκιο. Εγκρίνεται. Μετά την τροπολογία παριθμών 9 υπάρχει η τροπολογία μετά την παράγραφο 9, 14 της κυρίας Χίρς υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τηλεοπτική σκέψη α, τροπολογία παριθμών 1 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την CA, γάμα α, η τροπολογία 2 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται στο σύνολό τη τώρα η, ε, το σχέδιο γνωμοδοτήσεως το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Υψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 υπέρ. Δύο εποχές. Άρα εγκρίναμε τη γνωμοδότησή μας για τον προπολογισμό και προχωρούμε στο σημείο 5 της Μερσής εντάξεως. Έχουμε δηλαδή την εξέταση του σχεδίου ε, επιστολής ε, σχετικά με την γνωμοδότηση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης στο πλαίσιο της υπόθεσης ΛΙΝΑΚ που έχει ε, εκκινήσει η κυβέρνηση της Δανίας, η υπόθεση της κυβέρνησης της Δανίας. Για να δούμε λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά έχουμε γνωμοδότηση για την υπόθεση της, του ομίλου Ντάνφος, πάλι από τη Δανία, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ποιος είναι υπέρ της επιστολής. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και εν τέλει έχουμε ένα θέμα κλώστο υφαντουργικό σχετικό με τη Γαλλικία, κυβέρνηση της Ισπανίας αυτή τη φορά, πάλι κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η αρχική επιστολή όμως πρέπει να σας πω, η επιστολή που έχει διανεμηθεί δηλαδή, ε, εμπεριέχει ένα σφάλμα. Στην τρίτη παράγραφο, στο αρχικό κείμενο, δεν υπάρχει διαγραφεί. Δεν έχει απαλληφθεί δηλαδή η παράγραφος. Απλώς στόχος ήταν η παριθμόν τέσσερα παράγραφος Donc vous avez, vous avez dans vos dossiers, vous avez sur vos, vos tablettes Λοιπόν, θα το έχετε δει, ξαναρχίζει ο Πρόεδρος, ε, υπάρχει το διορθωμένο κείμενο στους φακέλους σας. Εάν δεν έχετε κάποια δυσκολία εσείς ε, κατανόησης ή αντίρρηση κτλ, ψηφίζουμε ακριβώς αυτή την έκδοση που είδατε. Δηλαδή, στην πρώτη παράγραφο συμφωνούμε με την Επιτροπή και την πρότασή της, στη δεύτερη εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την προαγωγή της κινητικότητας, Στην τρίτη εκφράζουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέτρα υποστήριξης, βελτίωσης των συνθήκων εργασίας και ε, προσωπικού βίου με τα 400 ευρώ και στο τέταρτο εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι περίπου το 50% των μέτρων για την κατάρτιση και την μάθηση ε, δεν ε, θα είναι αυτά που θέλαμε. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν, δεν υπάρχει αντίρρηση πολύ καλά. Ψηφίζουμε το, την επιστολή τη σχετική με το αίτημα της Ισπανικής κυβερνήσεως, παρακαλώ, στο κείμενο που είδατε, υπέρ, κατά, αποχές. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας και προτείνω αμέσως να περάσουμε στο σημείο 8 την εξέταση δηλαδή σχεδίου γνωμοδοτήσεως την οποία έχουμε αναλάβει προς την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ για την εφαρμογή της οδηγίας περί Η κατουσία ουσίαν αρμόδια ε, για την έκθεση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι η κυρία Γκέπχαρτ και για μας συντάκτης νομοδότης ο κύριος Μπενάμιας, τον οποίο δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Θα έλεγα ε, οδηγία περί υπηρεσιών υπαριθμών 2, η επιστροφή. Έχουμε πολλές συζητήσεις λοιπόν Διεξαγαγή, πολλοί άριθμες συζητήσεις. Καταφέραμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ίδια επί ε, συντάκτρια τη εκθέσεω, την κυρία Γκέπχαρτ δηλαδή, φτάσαμε σε συμβαστική λύση. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα τώρα, έστω και αν κάποια κράτη δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στις λύσεις που θέλαμε ως προς την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η γνωμοδότηση είναι σύντομη, όπως ορίζουν οι κανόνες του Κοινοβουλίου, μόνο 500 ίσου χαρακτήρες δηλαδή, παρά τη σημασία και την έκθεση τη οδική περιπτώσεων. Εν πάση περιπτώσει. Η ιστορική αγορά των υπηρεσιών, λέμε, θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρω με την ταυτόχρονη διαφύλαξη και του κοινωνικού μοντέλου τη Ευρώπης. Αυτονόητο. Επίσης λέμε ότι θα, έχουν, θα πρέπει να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη θέσεων εργασία ε, αυτές οι διατάξεις, βασικό ρόλο δηλαδή της οδηγίας, μάλλον της έκθεσης αυτής ορίζουμε την εξέταση της εφαρμογής οδηγίας και την, ε, τον αντίκτυπό της ως προς την ε, απασχόληση και την ασφάλεια. Επίσης, καθώς από την έξοδο οδηγίας έχει τεθεί και σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, επισημένω, χωρίς σου υπερβολικές ε, λεπτομέρειες, σε διάφορα σημεία 3, 9, 14, τα άρθρα της συνθήκης δηλαδή ε, ή το πρωτόκολλο 26 που ακριβώς παραπέμπουν στη σχετική οδηγία, στην οδηγία της σχετικής υπηρεσίας. Επεκτείνεται επίσης το πεδίο εφαρμογής ε, στις Υπηρεσίε γενικού συμφέροντος, υπηρεσίε υγεία περισσότερες εκ των κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί υπήρχαν κάποιες γκρίζες ζώνες. Και επίσης επισημαίνουμε ρητά ότι δεν αφορά το εργατικό δίκαιο ούτε την νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση που ισχύει στα κράτη-μέλη. Και για μένα είναι σημαντικά είναι η παράγραφος αυτή. Αυτό που δεν βλέπουμε λοιπόν ακόμα τουλάχιστον, είναι η οδηγία εκείνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εξηγεί πραγματικά τι σημαίνει η υπηρεσία γενικού συμφέροντος. Ποια είναι εκείνη η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή ποια δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ποια είναι πραγματικά οικονομικού χαρακτήρα, καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου τι είδους δικαιώματα μπορούν να αντλήσουν από την έννοια αυτής της υπηρεσίας γενικού συμφέροντος ε, τα κράτη-μέλη. Επίση, η έννοια τη ενιαία θηρίδα δεν έχει προχωρήσει σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητη όμω για την ε, ικανοποίηση αυτών των όρων τη οδηγία. και γι' αυτό κάνουμε τη σχετική παραπομπή και στο άρθρο τη συνθήκη για την περιοδική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα τη εφαρμογή οδηγία, για την απασχόληση τη ποσοτική από και ποιοτική πλευρά, Στο άρθρο 150 συγκεκριμένα τη συνθήκη τη Ρώνης, της Λισαβόνα. και γι' αυτό λοιπόν λέμε ε, ότι πρέπει να περάσουν οι συμβαστικές λύσεις οι οποίες είχαμε ε, στο παρελθόν το έχουμε συμφωνήσει αυτό και άλλωστε έχουμε προχωρήσει συνεργασία με την κυρία Γκέπχαρτ ε, τα διάφορα οι διάφορες δυνατότητες προνόμια και μέτρα υπέρ των πολιτών που ισχύουν ήδη θα πρέπει να ακυρωθούν ή να ματαιωθούν και γι' αυτό θα σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την απομόνωση. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτή τη θαυμάσια εργασία και το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα όλα αυτά να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και η ομάδα μου θα καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για θέματα ευαίσθητα και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι στο σημείο 4 λέει ο εισηγητής ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια οδηγία η οποία θα διασαφηνίζει τις ε, διάφορες έννοιες εμπορικέ δηλαδή υπηρεσίε, υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο κτλ. Και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη την κατάσταση που αφορά στι διάφορε χώρε μελίου όσον αφορά την εφαρμογή αυτή τη οδηγία πράγματι δεν έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες μέλη την οδηγία αυτή. Οπότε θα ήταν σημαντικό να προσθέσουμε ότι υπάρχουν 12 χώρες μέλη οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει την οδηγία με τρόπο ολοκληρωμένο. Αυτό νομίζω ότι είναι απαράδεικτο για τους πολίτες των χωρών μελών, όπως επίσης και για τους πολίτες των χωρών μελών που έχουν εφαρμόσει την οδηγία αυτή. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει μια ομοιογένεια και οι χώρες που έχουν σημείωση καθυστέρηση να την καλύψουν. Σημείο 5. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια προσθήκη. Όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία θηρίδα η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για να απαντήσει στα ερωτήματα και για να πληροφορεί τους πολίτες. Και να πω επίσης ότι είμαι υπέρ του σημείου 6 του που ζητάει μια περιοδική έκθεση όμως και εδώ πάλι θα πρότεινα να κάνουμε την παράγραφο αυτή πιο καθοριστική πιο σημαντική δηλαδή να λέμε ότι θα πρέπει η έκθεση αυτή να είναι τουλάχιστον ετήσια και η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιγράφει την κατάσταση που αφορά όλες τις 27 χώρες μέλη ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες σύγκρισεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Τουρινέν και μετά η κυρία Μάρκιν, κυρία Τουρινέν. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω δανέζικα και θα μιλήσω σιγά, αργά. Παρακολουθώ το φάκελο αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον και πριν γίνω ευρωβουλευτής να πω ότι το, θέμα αυτό ήταν μια από τις πιο σημαντικές συζητήσεις που αφορούσε όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους δηλαδή η οδηγία για τις υπηρεσίες και επιπτώσεις, του, επιπτώσεις της στον κόσμο της εργασίας από νεαρά ηλικία λοιπόν παρακολουθώ τις επιπτώσεις αυτής της οδηγίας οπότε να πω ότι σχετικά με την εφαρμογή το σχέδιο γνωμοδότησης αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι θαυμάσιο μάλιστα, σε σχέση με τα αιτήματα που προβάλλει και το περιεχόμενό του. Και υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία εμείς ως ομάδα θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε. Όμως και η Επιτροπή Απασχόλησης, δηλαδή εμείς εδώ ως Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να επαληθεύσουμε τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο όσον αφορά την απασχόληση. Αυτό ακριβώς νομίζω να λείπει στο σχέδιο της γνωμοδότησης, δηλαδή ο εντοπισμός των πραγματικών προβλημάτων. Γιατί το θέμα εδώ δεν έχει να κάνει και τόσο με την οδηγία για τις υπηρεσίες πέραν κάποιων πτυχών νομικών εφαρμογής οδηγίας σε κάποιες χώρες μέλη. Το πραγματικό πρόβλημα αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν εκτός συνόρων μέσω συμβάσεων. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε, μάλλον να υπενθυμίσουμε ότι και αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανταχθούν σε αυτή την οδηγία και νομίζω αυτός ακριβώς ο κρίκος λείπει στην αλυσίδα. Η άλλη πτυχή που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, όπως είπαν και οι σοσιαλδημοκράτες, νομίζω θα πρέπει να κάνουμε πιο σαφή την παράγραφο 5, 6 θέλει να πει η ομιλήτρια, για τις περιοδικές εκθέσεις. Και όπως έλεγε και η συνάδελφος προηγουμένως, η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια, ώστε να συζητά την κατάσταση σε όλες τις χώρες μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και την απασχόληση. Και μετά έχουμε και άλλο ένα μεγάλο δίλημα όταν μιλάμε για τον ορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλεια. Καταλαβαίνω υπάρχει κάποια σύγχυση εδώ, αλλά αυτή η παράγραφος, να πω την αλήθεια, με ανησυχεί λιγάκι, γιατί φαίνεται ότι ο Μισελ Μπαρνιέ ανέφερε το ενδεχόμενο ομοιογενεοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει, τι θα υποβάλει συγκεκριμένα ω προτάσει ο, ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Όμως ο τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό. Και το γεγονό ότι θα έπρεπε να παρουσιάσουμε, να υποβάλουμε μάλλον ένα ορισμό θα ήταν καλό. Το κακό θα ήταν να υποβάλουμε ως πρόταση έναν ορισμό ο οποίος θα ήταν περιοριστικός και θα άφηνε καθόλου περιθώρια όσον αφορά τις χώρες μέλη για να περιλάβουν ακριβώς αυτές τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες. Και να πω ότι συμφωνώ με αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση και βεβαίω θα πρέπει να δούμε ακριβώ να δούμε ποιε είναι οι προθέσει τη Κομισιόν. Συνοψίζοντα λοιπόν, θα πρέπει να περιλάβουμε του εργαζομένου εκτό συνόρων που είναι ένα πρόβλημα συγκεκριμένα που θα πρέπει να λυθεί. Θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει μια αξιολόγηση πιο ισχυρή εκ μέρους της Κομισιόν και τρίτον θα πρέπει να ορίσουμε σωστά τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στο σημείο 4. Και εδώ ως πράσινοι θέλουμε να είμαστε έτσι πιο σαφείς. Και κάτι το τελευταίο. Ως μέλος της ομάδας της Επιτροπής μάλλον ΙΜΚΟ Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η δική μας Επιτροπή να έχει μια θέση ξεκάθαρη. Έχω την εντύπωση ότι δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία στις χρηματοοικονομικές προοπτικές. Είναι λοιπόν σημαντικό εμείς να αναφέρουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι επιπτώσεις της οδηγίας αυτής για τους εργαζόμενους. Αυτά θα πω και σας ευχαριστώ για αυτή την πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ Άρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε στην γνωμοδότηση. Καταρχήν μια, ένα γενικό σχόλιο. Νομίζω ότι θα ήταν θετικότερο για την οδηγία και όπως είπαν διάφοροι σχολιαστές χρειαζόμαστε μια γενική εφαρμογή σε όλε τι χώρε αυτής τη οδηγία, υπάρχουν χώρε που δεν την έχουν εφαρμόσει και νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο σημείο εδώ τουλάχιστον όσον αφορά βεβαίω και την τωρινή οικονομική κρίση. Σε σχέση με το σημείο 2 θα συμφωνούσα ότι υπό το φως της νέας συνθήκης χρειαζόμαστε μια νέα ερμηνεία για, κάποιους, για, για κάποια άρθρα και συμφωνώ με αυτή την άποψη Κάτι άλλο, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια σημεία σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία Ίσως ο Ζαν θα μπορούσε να αναλύσει περισσότερο κάποια από αυτά τα σημεία ώστε να έχουμε εμεί μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι έχει κατά νου και να δούμε ακριβώ τι επιπτώσει έχουν αυτέ οι παράγραφοι. Θέλουμε λοιπόν κάποιε παραπάνω πληροφορίε για το τι έχει κατά νου εδώ και επίση καταγράφω το σχόλιο τη πράσινη συναδέλφου προηγουμένω που έλεγε για το ενδεχόμενο κάποιοι ορισμοί να είναι ίσω υπερβολικά περιοριστικοί είναι σαφές εδώ ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέμε, τι εννοούμε. Μετά, για το σημείο επαφή να πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες μου από το Συμβουλίο Ανταγωνιστικότητας πριν από ένα χρόνο μου λένε ότι οι χώρες μέλη δεν έχουν εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμόσουν και να πω ότι συμφωνώ με την ιδέα του ο, του ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται στο εξωτερικό. Τέλος, να πω ότι ρίχνοντα μια ματιά και ποιοτική και ποσοτική όσον αφορά την απασχόληση, την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο μιλούσαμε για τις επιπτώσεις της οδηγίας αυτής και την στάση του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Να ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά για αυτή την γνωμοδότηση και να πω ότι συμφωνώ απόλυτα όλα σε επενπρολύσαντες ίσως ενδεχομένω να πρέπει να κάνουμε κάποιε μικρές αλλαγές. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, άλλωστε συμφωνώ με τους συναδέλφους μου. Θα ήθελα περισσότερο να επικεντρωθώ στο σημείο 4 θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες ε, πάρα πολλές περιπτώσεις αποτελεί ουσιαστικά μια οδηγία ορόσημο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να επιβάλλει τη δική του άποψη στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γιατί θα θυμάστε ότι διαφωνήσαμε με την αρχή της χώρας προέλευσης και τελικά πέρασε η δική μας η άποψη, η δική μας η θέση μέσα από τις καταπληκτικές βέβαια προσπάθειες που έκανε η κυρία Γκέπχαρτ. Το λέω αυτό γιατί νομίζω θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Οι τομείς που έχουν μείνει εκτός οδηγίας είναι τομεί όπου ο ίδιος ο πολίτης, όχι μόνο το κοινοβούλιο, ο ίδιος ο πολίτης είχε εκφράσει ανησυχίες. Δεν ήθελε να δει τους κοινωνικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθοδηγούνται μόνο από υπολογισμού, από συμφέροντα οικονομικά στα πλαίσια της αγοράς δηλαδή. Και είναι σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να δούμε πώ εφαρμόζεται η οδηγία αυτή, το οποίο βέβαια είναι δύσκολο γιατί 12 κράτη-μέλη δεν την έχουν ακόμα εφαρμόσει. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώ λειτουργεί η οδηγία αυτή στην πράξη. Όσον αφορά τώρα το σημείο 4, ο συγητής για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίες Επιτροπής μας για το μέλλον των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος θα ήθελα να εκφράσω λοιπόν την άποψή μου και ελπίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση μέχρι τα τέλη του έτου. Πάντω, η Βελγική Προεδρία οργανώνει ένα φόρουμ στα τέλη Οκτωβρίου για τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο και νομίζω ότι ε, θα είναι ένα φόρουμ ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα θέσει ουσιαστικά τι βασικέ προτεραιότητε στον τομέα αυτό για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το εξή ότι από τη στιγμή που εγκρίθηκε η ε, οδηγία αυτή, εγκρίθηκε στη συνέχεια από όλα τα κράτη-μέλη και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και όπως λέει και ο συντάκτης της ε, νομοδότησης ε, περιλαμβάνει και το άρθρο 14, που αναφέρεται σε νομικές διατάξεις όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινή ωφελία και τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή λοιπόν της οδηγίας θα πρέπει να αναφέρεται περισσότερο και στο άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει απαραίτητη αυτή η διόρθωση. Και μια τέτοια εφαρμογή βέβαια του άρθρου αυτού και βάσει των όσων θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν θα περιορίζει τις εθνικές αρμοδιότητες, αρμοδιότητες δηλαδή των κρατών μελών όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Για τις υπηρεσίες αυτές τελευταία ανάλυση τα κράτη-μέλη είναι άμεσα αρμόδια. Τουλάχιστον όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θέσει ένα πλαίσιο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο και υπηρεσιών κοινή ωφελία. Είναι πολύ σημαντικό να φερόμαστε επίση και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώ επίση και στο πρωτόκολλο υπαριθμών 26, καθώ ε, και ο χάρτη και το πρωτόκολλο αναφέρονται στι υπηρεσίε αυτέ. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική σε σχέση βέβαια με αυτό το οποίο επιτύχαμε πριν από μερικά χρόνια για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ο... Η σημερινή μορφή της οδηγίας αυτής και οι σημερινές ε, παρεκκλήσεις από την οδηγία αυτή οφείλονται ουσιαστικά στις ισχυρές αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το τελικά καταφέραμε να περάσουμε τη δική μας θέση Και βέβαια δεν θα πρέπει να, θεωρώ να αναφερθώ μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία στη συνέχεια ενέκριναν με τη σειρά του και τη συνθήκη τη Λαβόνα. Επομένω, δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι και τα εθνικά κοινοβούλια που ζητούν να εφαρμοστεί η οριζόντια κοινωνική ρήτρα του άρθρου 9 τη συνθήκη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι η οδηγία για τι υπηρεσίε εγκρίθηκε πριν να τεθεί σε εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα και αυτή τη στιγμή σε αξιολογούμε την εφαρμογή τη οδηγία αυτή θα πρέπει να συμπαραδειχθούν οι κοινέ ρήτρε που φέρνει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα πρέπει να σα πω επίση ότι οι υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια της δεύτερης ολομέλειας ε, του Σεπτεμβρίου. Θα ήταν ε, καλό να ζητήσουμε από τον Επίτροπο Άντορ αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια task force ε, υψηλού επίπεδου αντίστοιχη με αυτήν που είχε δημιουργηθεί για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, προκειμένου να δούμε τελικά αν μπορεί να βρεθεί ένα σημείο σύγκληση, ένα σημείο συμφιλίωση, συμβιβασμού, ανάμεσα στην νομική βάση για την εσωτερική αγορά και τις κοινωνικές ανησυχίες και κοινωνικές πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν μπορούμε επίσης να λάβουμε υπόψη μας και την, το ρόλο που διδραματίζουν ε, οι ε, τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και άλλες εθνικές ε, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές υπηρεσίες που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να συντονίζει τη δράση όλων αυτών των φορέων και που να μπορεί να επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ τους θα ήταν σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε την ιδέα αυτή προς τον Επίτροπο και θα ήθελα και τη δική σα υποστήριξη. Μπορώ να σας δώσω μάλιστα και ένα αντίτυπο του εγγράφου που θα ήθελα να υποβάλω στην Ολομέλεια. Η κυρία Φιγκερέντο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορούσα νομίζω να πω Πρόεδρε για το θέμα αυτό το εξής. Οι καθυστερήσεις είναι βέβαια αρνητικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Επειδή ενδεχομένω θα υπάρξουν χώρες οι οποίες θα παρουσιάζουν περίπλοκες καταστάσεις, κοινωνικές δηλαδή και οικονομικές, όπου μια απελευθέρωση, όπως προβλέπει η οδηγία, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιδίνωση της ανεργίας Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αμφιβολίες σε σχέση με την κατάσταση που αφορά την έλλειψη εφαρμογής οδηγίας των 12 χώρες μέλη. Αυτό σημαίνει βεβαίως τώρα ότι θα πρέπει να έχουμε ιδέες ξεκάθαρες για να δούμε ακριβώς ποια επιχειρήματα έχουν υιοθετήσει οι διάφορες χώρες μέλη ώστε να κάνουμε μια μελέτη αντίκτυπου της εφαρμογής της οδηγίας αυτής στις χώρες όπου ήδη έχει εφαρμοστεί. Κατά την άποψή μου η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα γιατί θα εξαρτηθεί ακριβώς από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ αρνητικό σε κάποιες χώρες μέλη παρά τις τροποποιήσεις που έκανε το Κοινοβούλιο και υπό το φως των απόψεων, των εκδηλώσεων και των διαδηλώσεων που είχαμε ακριβώς μπροστά από το κτίριο του Στρασβούργου κιόλας. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι έχω κάποιες ανησυχίες σχετικά με τις πιο προβληματικές πτυχές της υπόθεσης αυτής. Δηλαδή, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε τη διευκρίνηση των ορίων της οδηγίας. Εγώ νομίζω ότι αυτές είναι δυσκολίες οι οποίες θα μπορούσαν να εμφανιστούν στους τομείς αυτούς και συμφωνώ με τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο εισηγητής. Τελικά να πω ότι θεωρώ πως είναι σημαντικό να έχουμε να εχουμε έχουμε μία μελέτη ξεκάθαρη, ένα follow-up που να παρουσιάζει την κατάσταση που έχει, ώστε να προσπαθήσουμε μετά να διατυπώσουμε ή να επαναδιατυπώσουμε ε, γνώμες και απόψεις για την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. κυρία Σλοβισκά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ε, συζήτηση για την οδηγία περί υπηρεσιών συζητούμε συχνά την αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών πτυχών. Αν όμως πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση, θα πρέπει πιστεύω να υιοθετήσουμε πολύ σαφή κριτήρια με στοιχεία εξάντε, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, αμφιβολίες προς την Γιατί όταν ε, έγινε η επεξεργασία αυτών των στοιχείων για την οδηγία στι χώρες μας, οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι τώρα. Και θέλω επίση να πω ότι η Επιτροπή ΕΜΚΟ έχει προβλέψει για τις 29 Σεπτεμβρίου τη διεξαγωγή ε, συζητήσεως σε εργαστήριο όπου θα παρουσιαστούν τα πορίσματα από την εφαρμογή της οδηγίας στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία ανάλυση την οποία ανέλαβε ανεξάρτητη ε, επιχείρηση, εταιρεία. Η δε γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟΠΟΤΗ κατάλαβα πρόκειται να στηριχθούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρότεινα να αναφερθεί η λήψη αποφάσεων στην γνωμοδότησή μας. Η Πρόεδρος. Ναι, εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ καταρχάς ε, τον εισηγητή για την ε, σύμβαση για την συμβολή του στην ε, δουλειά αυτή. Ξέρουμε βεβαίως ότι όταν κανείς έχει γνωμοδότηση σε τόσο περίπλοκα θέματα υπάρχουν περιορισμοί. που μπορεί να καταστάσουν το έργο μας πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει όμως και πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 1 ως προς την ανάλυση σχετική με την οδηγία και της, ε, τη συμβολή της στην, ε, δημιουργία θέσεων εργασία. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να την κοιτάξουμε με μια κάποια ε, προσοχή και να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα διατυπώσουμε αυτά τα συμπεράσματα, διότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με κάθε είδους θέση εργασίας που δημιουργείται Θέλουμε συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς, θέλουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας. Και μην ξεχνάτε ότι όταν, ε, επεξεργαστήκαμε, όταν είχαμε την επεξεργασία της οδηγίας, ένα από τα κύρια ζητήματα πάνω στα οποία κρίθηκε και η μοίρα της οδηγίας ήταν να μην δημιουργηθούν, ε, να μην τίνουμε προς ε, αβέβαιες ή πολύ σύντομης ή πολύ κακών συνθήκων ε, θέσεις εργασίας. Αυτό λοιπόν νομίζω θα πρέπει να το ε, υπογραμμίσουμε μέσα από τους όρους που ορίζει και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με την έννοια και της βιώσιμης θέσης εργασίας που θα πρέπει να συμπληρώσουμε και την, ε, το θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας το οποίο θα πρέπει να περιγράφουμε μέσα από τις προϋποθέσεις και αυτές βέβαια που ορίζει η ίδια η οδηγία αλλά και εκείνες ε, από τις οποίες η τελευταία ανάλυση εξαρτάται και η εφαρμογή υλοποίησης οδηγίας στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε και τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να ε, αξιολογήσουν τις ε, εκτελήξεις αυτή τη στιγμή. Και επίσης, θα πρέπει πιστεύω να συζητήσουμε και πάλι το τι διακυβεύεται με την προοπτική της ξένασης της νέας συζήτησης της οδηγίας για την απόσπαση εργοζομένων, που ξέρω ότι ανησυχεί πολλούς από εμάς εδώ. Και αυτές είναι οι προτάσεις που θέλω να διατυπώσω. Εάν υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Όχι από ό,τι φαίνεται. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μάρτεν Πράτ, Μάρτ από την Κομισιόν, αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, στα αγγλικά. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνετε στην Επιτροπή να λάβει το λόγο. Να ευχαριστώ τον κύριο Μπεναμιάς, τον εισηγητή, για το σχέδιο. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι η Επιτροπή Θεωρείται σημαντικό το ότι μπορεί να στηρίζεται στην ε, στήριξη του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής σας, δηλαδή την ε, πίεση μπορείτε να ασκήσετε στα κράτη-μέλη, ε, ιδιαίτερα για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Έχουμε διαξεχάγει διαπραγματεύσεις σκληρές και δύσκολες. Πιστεύουμε ότι το να εφαρμοστεί ορθά η οδηγία από τα κράτη-μέλη θα είναι εις όφελος και των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ε, γνωρίζετε βέβαια τα στοιχεία, τα αριθμητικά. Γνωρίζετε πολύ ε, καλά όλοι σας ότι το 75% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εξασφαλίζει ο τομέας των υπηρεσιών και τεράστιο ποσοστό επίσης από την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τον τομέα των υπηρεσιών. Ξέρετε επίσης ότι η τάση τα τελευταία χρόνια ήταν ο καθαρός ε, το καθαρό ισοζύγιο υπέρ της δημιουργίας της εργασίας να προέρχεται από τον ίδιο αυτό το τομέα των ε, υπηρεσιών και με την τρέχουσα οικονομική κρίση διαπιστώνεται ότι αυτός ακριβώς ο τομέας των υπηρεσιών είναι εκείνο που μπορεί να αντισταθεί περισσότερο στον αντίτυπο στις επιπτώσεις της κρίσης. Άρα πρέπει ιδιαίτερα να τον διαφυλάξουμε και αυτό όπω είπα προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πολίτη ο οποίος αποφέλεται των υπηρεσιών ή εργάζεται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Πολλοί εξημών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το, την πρόοδος προς την υλοποίηση της οδηγίας και ο εισηγητής ο κ. Μπεναμιάς και ο κ. Κρίστενσεν, η κ. Χάκιν, ο κ. Ντερόσα εξέφρασαν αντίστοιχες ανησυχίες στι παρεμβάσεις τους. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις προς την ε, ε, εφαρμογή, την υλοποίηση τη οδηγία από τα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν σημαντικέ πρόοδοι τελευταία, τις οποίες πιστεύω οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό και στην πίεση που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο, το οποίο σε επίπεδο Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα, αλλά και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει διατηρήσει την πίεση για τα κράτη-μέλη και βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσά λέει του βουλευτέ που ασκείτε πίεση στα κράτη-μέλη, τη κυβέρνηση τα στοιχεία τα αριθμητικά τα οποία ακούστηκαν ε, από ορισμένε παρεμβάσει ότι 12 κρατημέλη ακόμη δεν εφαρμόζουν την οδηγία δεν ισχύουν πλέον. Είναι περίπλοκο βέβαια το ζήτημα τη υλοποίηση καθώ πρόκειται για μια δέσμη μέτρων. Πολλά πράγματα μένουν να γίνουν. Αλλά για να σα δώσω μια ιδέα του πού βρισκόμαστε ω προ τα κύρια ζητήματα τη οδηγία. Οριζόντια νομοθεσία λοιπόν υλοποιούν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή τη οδηγία αυτό είναι το σύστημα, εκτό και να αποφασίσουν να προχωρήσουν με χωριστά νομοθετικά κείμενα ε, κατά περίσταση. Εδώ έχουμε λοιπόν 25 κράτη-μέλη τα οποία έχουν ολοκληρώσει το, την οριζόντια νομοθεσία. Μόνο δύο είναι τα κράτη στα οποία εκκρεμεί ακόμη αυτό το νομοθετικό έργο. Διορθώνω, λέει ο Μιλήτρια, 24 ακόμα είναι τρία τα κράτη δηλαδή, τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο διατύπωση ή σχεδιασμού τη νομοθεσία, τη οριζόντια νομοθεσία. Ω προ τι τροποποιήσει τώρα, τι μεταρρυθμίσει που θα πρέπει να εισαχθούν όχι μόνο σε επίπεδο οριζόντια νομοθεσία, αλλά και στην προσαρμογή, την απλούστευση, την άρση των όποιων φραγμών ή σε υφιστάμενα νομοθετικά έργα. Έχουμε 21 εκ των 27 κράτη-μέλη που έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά στο πεδίο αυτό. Βέβαια, αυτό λαμβανομένου υπόψη και του όγκου που προκύπτει ω προ την ανάγκη τα κράτη-μέλη να ε, προβούν σχετικέ νομοθετικέ μεταρρυθμίσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 100 ίσω νομοθετήματα ανά κράτο μέλο και χωρί να θέλουμε να ε, κολακεύουμε τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ως Επιτροπή ότι μπορούμε να έχουμε με λίγη ακόμη πίεση πολύ καλά και ικανοποιητικά αποτελέσματα ταχύτατα. Τα σημεία ε, η μονοθυριδική επικοινωνία, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλα τα κράτη-μέλη. Η μονοθυριδική προσέγγιση λοιπόν είναι ουσιαστικά αυτά τα κέντρα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως θα τα λέγαμε, που θα επιτρέπουν στον πολίτη όχι μόνο να λαμβάνει ενημέρωση αλλά και να ε, διεκπεραιώνει ζητήματα σχετικά με τη δημόσια διοίκηση Αυτά έχουν πάλι προχωρήσει στα περισσότερα εκ των κρατών μελών. Και πάλι δεν επαναπαυόμεθα ω Επιτροπή. Δεν θεωρούμε ότι έχει λήξει το ζήτημα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον. Α, πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση και να εξηγήσουμε στα κρατη μερα ότι χρειάζεται να ολοκληρώσουν αυτήν την καλή δουλειά. Αλλά είναι σημαντικό ταυτόχρονα να πούμε ότι είναι πολλέ οι προσπάθειε των κρατών μελών και σημαντική η πρόοδο που έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ασήμαντη. Επίση, επιτρέψτε μου, σε ένα ζήτημα να επισημάνω ότι στην υλοποίηση αυτή την οποία έχουμε παρακολουθήσει σχέση με τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι ήταν γενικά πολύ θετικό το κλίμα ως προς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Δηλαδή και οι κυβερνήσεις υπέβαλαν τις προτάσεις τους και τα κοινοβούλια συζήτησαν χωρίς αντιδράσεις ήταν γενικά θετικό το κλίμα για το πεδίο εφαρμογής. Για τον κύριο Μπεναμιάς και τη μονοθυριδική προσέγγιση ε, και βέβαια την προσέγγιση στα άλλα ζητήματα, η Επιτροπή θα συμφωνήσει με τη θέση του συντάκτη, της νομοδότηση, αλλά πιστεύω ότι είναι δεδομένο ότι άπαξ και τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι ενιαίε θηρίδες δεν τίθεται πλέον ζήτημα του ε, να καταστούν υποχρεωτικέ σημεί. Δεν θα συζητηθεί πλέον θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ σημεί. Γιατί θα δουν οι κυβερνήσει, τα κράτη, ότι μπορούν να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή σε μικρομεσαίες επιχειρήσει που θα οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασία κτλ. Και δεν βλέπω κανέναν να λέει Α, όχι, δεν θα το κάνω. Φερρυπίν τα φορολογικά. Ένα παράδειγμα. Τα φορολογικά συστήματα δεν καλύπτονται από την, υπηρεσία, από την οδηγία περί υπηρεσιών. Ναι, αλλά μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να συσταθεί, ένα επιχειρηματή που θέλει να φτιάξει μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα χρειαστεί και συμβουλέ στον τομέα αυτών. Επομένω, θα πρέπει να προσφερθούν και αναλόγω θα πρέπει να γίνει προσαρμογή στην εθνική νομοθεσία εκ των πραγμάτων. Είναι λοιπόν επιθυμητό να προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες ή πληροφορίε σε αυτές τι ενιαίες και επίσης ο αντίκτυπος στην απασχόληση, ιδιαίτερα όπως είπατε ποιοτικέ θέσεις εργασίας μέσα από την οδηγία, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Ένα ακόμα ίσως θα πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι πρέπει να προβλέψουμε επαρκή χρόνο για τις δομικές αλλαγές, την προσαρμογή δηλαδή των κρατών μελών που αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά μέσα στην νομοθεσία και από εκείνη τη στιγμή και μετά να περιμένουμε να δούμε τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Δεν θα αλλάξει δηλαδή τίποτα στην πραγματική οικονομία μόνο και μόνο γιατί άλλαξε ένας νόμος. Πρέπει να αλλάξουν σιγά σιγά και οι, νομο... και οι νοοτροπίες, ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο. Οι αναθεωρήσεις, οι μεταρρυθμίσεις αυτές και μόνο δεν μπορούν να φέρουν το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ίσως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο έτσι ώστε να δούμε, να περιμένουμε να δούμε και τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέση σε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σα ενδιαφέρει για, το, για την πρόοδο στην υλοποίηση αυτή τη οδηγία. Έχουμε τη σχετική προσαρμογή ε, από το τελευταίο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται να γίνεται τακτικά αυτή η ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας, αλλά αν του μεταξύ θέλετε κάποια άλλα στοιχεία, είμαστε στη θέση σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι, κύριε Μπάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν είπε ότι σε 24 χώρες έχει ολοκληρωθεί η νομοθεσία σε 12 δεν εφαρμόστηκε, αλλά το θέμα είναι ότι το πιο πρόσφατο έγγραφο που διάβασα ήταν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βεβαίω θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στην Επιτροπή και δεν ξέρω τι χρονοδιάγραμμα έχουμε, αλλά θα υποστηρίξω το αίτημα της συναντέλφου στην ακρόαση στο τέλος του μήνα να μας ενημερώσετε και θα ήθελα κάποιες εδώ κατευθύνσεις κάποια καθοδήγηση από το Προεδρείο αλλά τέλο πάντων συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση τη αδέλφου. Ο εισηγητή. Εμένα αναφέρατε. Α, συγγνώμη δεν άκουσα καλά. Ωραία. Ε, ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν το λόγο. Πρόεδρε, είπατε κι εσείς ότι έστω και θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα ξέρουμε ότι αυτή η οδηγία αφορά κάποια πράγματα που ποικίλουν που έχουν ποικιλομορφία και από την αρχή που συζητήθηκε η οδηγία αυτή στο Κοινοβούλιο δεν είδα σημαντικές αντιρρήσεις από τους παρεμβαίνοντες. Εγώ είμαι πάντως διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας με συγκεκριμένο τρόπο και βεβαίως να ξέρετε ότι η Επιτροπή μας δεν θα υποκαθιστήσει, υποκαταστήσει την κυρία Γκέπχαρτ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε αλλά να πω ότι ό,τι και να κάνουμε θα είναι θετικό. Να πω επίσης ότι η Κομισιόν ζητάει βοήθεια από το Κοινοβούλιο και εγώ με τη σειρά μου ζητώ βοήθεια από την Κομισιόν όταν έχουμε ένα θέμα που επανέρχεται στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές όπως ακριβώς είναι το 4 και εγώ βέβαια να βοηθήσω την Κομισιόν αν η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της Όταν μας λέτε ότι από τις ηγεσίε δεν τέχτηκαν πολλά ζητήματα, τότε συγγνώμη, αλλά ο, ο αριθμός των πιέσεων που δεχόμαστε από διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες μας λένε είμαστε εμείς μέσα στην οδηγία δεν είμαστε, όλα αυτά χρειάζονται περισσότερη διευκρίνηση. Πρόεδρε, δεν σε ποιο σημείο ήτανε. Αλλά τέλος πάντων ε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, χρειαζόμαστε βιώσιμη απασχόληση, απασχόληση που θα διαρκεί και όχι ότι να είναι. Για την κυρία του να πω ότι συμφωνώ μαζί της, διαφωνώ μόνο στο γεγονός ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε κοινωνικές πιέσεις. Όχι, αυτό αφορά άλλα θέματα, έστω και αν είπε η κυρία της Κομισιόν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί από την τελευταία έκθεση που είχαμε, ε, την έκθεση δηλαδή που δεχτήκα πριν ε, κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα για τους εργαζόμενους που εργάζονται στο εξωτερικό έστω και αν αυτό σχετίζεται άμεσα με την οδηγία για τις υπηρεσίες αφορά και άλλες οδηγίες ταυτόχρονα και έχουμε παρόμοιε περιπτώσει, βεβαίω όταν μιλάτε για σύγχυση, αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα που παρουσιάζει αυτή η οδηγία. Δηλαδή, τι σημαίνει ακριβώ μη οικονομική υπηρεσία κοινή ωφέλεια. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Δηλαδή, οι συνεταιρισμοί, τα διάφορα κοινοφελή ταμεία, όλα αυτά θα πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός. Βεβαίως υπάρχει κάποια έτσι δυσκολία ή είναι περίπλοκο το θέμα αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε την οικονομία της αγοράς με την κοινωνική οικονομία της αγοράς ώστε όλα αυτά να συνυπάρχουν. και είπε η Κομισιόν ότι στις υπηρεσίες υπάρχουν τομείς οι οποίοι άντεξαν στην κρίση, ξέρουμε αντίστοιχα ότι στον τομέα των συνεταιρισμών και των ε, οργανισμών κοινής ωφέλειας και σε αυτούς λοιπόν τους ε, τομείς η κρίση δεν ήταν και τόσο σοβαρή όσο στην παραδοσιακή οικονομία αγοράς ή στα άλλα συστήματα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά. Πάντως εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με όλους και θα ήθελα να πω ότι στην Επιτροπή μας όπως ακριβώς έγινε την προηγούμενη θητεία νομίζω καλύτερα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την κυρία Γκέπχαρτ στο να βρει ένα συμβασμό και να κάνει την οδηγία αυτή κάτι το οποίο πραγματικά θα βελτιώσει το σύλλογο των προοπτικών για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Τώρα θα πρέπει να καθορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα εξέτασης αυτής της νομοδότησης. Χρονοδιάγραμμα βεβαίως το οποίο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της πληροφορίας στην ΕΜΚΟ 30 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία οπότε εμεί θα ψηφίσουμε εδώ στις 8-9 ή του Νοέμβρη οπότε θα έχουμε το εξή χρονοδιάγραμμα κατάθεση τροπολογιών 27 Σεπτέμβρη μεσημέρι, εξέταση των τροπολογιών 25-26 Οκτώβρη και ψηφοφορία 8-9 Νοεμβρίου. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξή μας και περνάμε τώρα στο σημείο 10 που αφορά την πράσινη βίβλο για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιδοτικά συστήματα. Θα καλέσω την ομάδα του ΕΛΚ να μας μιλήσει η συγγήτριά τους δηλαδή για αυτό το σημείο. Θα ήθελα να τους δώσω το λόγο πρώτα, αλλά αφού αποσιάζουν θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Φίσερ ο οποίος θα μας παρουσιάσει εκ μέρους της Κομισιόν αυτή την πράσινη βίβλο. Και μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του ΑΣΑ. Κύριε Φυσέρα, έχετε λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου προσφέρει η Επιτροπή σας να σας παρουσιάσω την ε, πράσινη αυτή βίβλο. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο Και ελπίζω, ελπίζουμε ότι θα προκαλέξουμε ευρύτερο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά με την πράσινη βίβλο. Θα συνεχίσω τώρα στα αγγλικά, διότι έχω τις σημειώσεις μου στα αγγλικά, αλλά πολύ ευχαριστώ ότι έρθει η ώρα για τις ερωτήσεις να χρησιμοποιήσω και άλλες γλώσσες. Θα ξεκινήσω λέγοντας Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω πρώτα τις εξελίξεις από το τελευταίο συμβούλιο πριν από δύο ημέρες όπου παρουσιάστηκαν οι πολιτικές ε, για τα συνταξιδοτικά από τον Επίτροπο με την ανακοίνωση του 2011 του προγράμματος εργασίας που προβλέπει το 2011 λειτουργικές προτάσεις για την πολιτική που θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα και τη λειτουργία των στεξιωτικών συστημάτων. Θα θυμάστε επίσης ότι ο Πρόεδρος στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο το τελευταίο Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, είχε υπογραμμίσει τη σημασία των στεξιωτικών πολιτικών και μάλιστα έχει απαντήσει σε αντίστοιχα αιτήματα των βουλευτών. Έτσι λοιπόν η Πράσινη Βίβλος κινείται προς την υλοποίηση αυτών των λειτουργικών ιδεών, την εξασφάλιση πιο λειτουργικών, βιώσιμων, ασφαλών στρατιωτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου είναι ένα βήμα μεν η Πράσινη Βίβλος, όχι όμως ένα κείμενο συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων. Είναι απλώς ε, έναυσμα για συζήτηση. Το δεύτερο που περίμενε πιστεύω από μας ο Πρόεδρος της Επιτροπής εν προκειμένου ήταν να ξεπεράσουμε όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα τα όρια μέσα στα οποία συνήθως συζητούνται τα ζητήματα αυτά, τα λεγόμενα κουτιά, είτε είναι έκφυνη, είτε είναι Mark είτε είναι η Γενική Διεύθυνση για τα Κοινωνικά. Δηλαδή ο καθένας κοιτάει τα θέματα αυτά ανάλογα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δραστηριοτήτων του, ε, αλλά ταυτόχρονα δεν κοιτάμε, δεν κοιτούσαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα τις ε, συντάξεις ως συντάξεις, δηλαδή ως μια παροχή προς τον πολίτη, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει κάποια στοιχεία για να είναι ικανοποιητική. Αυτό λοιπόν ελπίζουμε ότι μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε με την πράσινη βίβλο, μία, όπως θα λέγαμε, ολιστική προσέγγιση, στο και κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει ολιστικός, μία σφαιρική προσέγγιση, για να το πω διαφορετικά, με τα εργαλεία, τα μέσα που έχουμε στη θέσή μας, που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα στοξιδοτικό, βιώσιμο, αηφόρο, λειτουργικό. Έτσι λοιπόν, ο δικό μου επίτροπο, ο κύριο Σάντερ, μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ και τον κύριο Ρεν, εκλήθησαν από τον Πρόεδρο. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι επίτροποι που έχουν στην αρμοδιότητά του θέματα συνταξιδοτική πολιτική. Αλλά οι τρει που σα προανέφερα είναι οι κύριοι ε, παράγοντε στην υπόθεση αυτή, οι πρωταγωνιστέ. έστω και να αναμειγνύονται κάποια άλλη επιτροπή ε, στι εργασίε αυτέ αυτές κατά καιρού. Βάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι έχω μια σφαιρική, ολιστική όπω λέγαμε προσέγγιση και αν επιτρέψετε πολύ σύντομα θα σα παρουσιάσω το έγγραφο και τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν, που καταγράφονται μάλλον σε αυτό. Στο πρώτο τμήμα εξετάζουμε το υπόβαθρο, τις τάσεις, τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα αυτή την εποχή. τρεις είναι, σε τρία στάδια θα έλεγα. Καταρχάς το ιστορικό, με δεδομένο και το παρελθόν των ιστορικών ε, ε, συστημάτων ε, που έχουν χαραχθεί, έχουν σχεδιαστεί σε μία περίοδο όπου το προσδόκιμο ζωής ήταν κάπου στα 60 έτη, ενώ τώρα έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής με αντίστοιχη μείωση της ε, ε, διάρκειας απασχόλησης λίγο πολύ, της προσδοκίας απασχόλησης. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν προχώρησαν σε μεταρρυθμίσει των του συστημάτων τα κράτη-μέλη, εν μέρη με σωστέ επιλογέ. Επίση βλέπουμε ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα ενδιαφέρει το κοινό, την, ε, τις δημογραφικές εξελίξεις που γνωρίζει πολύ καλά ως πρόβλημα το Κοινοβουλίο, γιατί έχει δει πολλές εκθέσεις στην υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, ανάλογα με το κράτος μέλος φυσικά αυτή η διάρκεια θα ποικίλει, η φυσική αναλογία μεταξύ εργατικού δυναμικού και συνταξιούχων ε, θα ανατραπεί αν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επαρκείς εργαζόμενοι, ότι θα, είναι, ότι θα δηλαδή, το εργατικό δυναμικό, γιατί εξελίσσεται η απασχολησιμότητα είτε των γυναικών είτε των μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει όμως η δημογραφία γενικά φέρνει κάποιες αλλαγές σημαντικές. Και επίσης βλέπουμε ότι αυτή η αυτές οι δημογραφικές εξελίξεις δρούν και λίγο ως κόδων κινδύνου, όπως θα λέγαμε, και για τα στοξιδοτοπικά συστήματα, γιατί θεωρούνταν ε, ότι το σύστημα χρηματοδότησης θα ήταν ε, μια διέξοδος για τα ευρωπαϊκά σταξιδοτικά συστήματα. Αποδεικνύεται όμως χάρη εντό εισαγωγικών στην οικονομική κρίση ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα τα ανταποδοτικά συστήματα έχουν τις ίδιες πιέσεις με τα μη ανταποδοτικά, άρα δεν αρκεί η ε, εξέταση της ε, δημογραφικής εξέλιξης και μόνο για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Και βλέπουμε ότι ιδιαίτερα σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα προβλήματα όπως η μακροχρόνια ανεργία μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές δυσκολίες γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς εισφορές για τη χρηματοδότηση των συντάξεων, δηλαδή της επιστροφής, της ανταπόδοσης, της λεγόμενης ανταπόδοσης. Επίσης κάτι που θα θέλω να υπογράψω ιδιαίτερο για την Επιτροπή σας και το είδαμε μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει η χώρα. Ορισμένα κρατημέρια δηλαδή ε, υιοθέτησαν ε, μεταρρυθμίσεις προσανατολισμένες προς την ε, βιωσιμότητα. Τα είδαμε αυτά και με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι ορισμένες ήταν πολύ θετικέ, αλλά οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό, είχαν σε μεγάλο βαθμό επίπτωση στις παροχές. Και αυτό μπορούμε να το δείξουμε και με, τις, με τους πίνακες που έχουμε ετοιμάσει. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή οδηγούν ουσιαστικά σε μια κατάσταση κατά την οποία για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έτη δηλαδή εισφορών μέσα σε ένα ταξιδιωτικό σύστημα α και με μια συγκεκριμένη ηλικία συνταξιοδότησης ε, οδηγούμεθα σε μια εξέλιξη κατά την οποία οι παροχές μειώνονται σημαντικά και πέφτουν ενδεχομένως κάτω από ένα όριο, το λεγόμενο όριο της καταλληλότητας, της επάρκειας δηλαδή, το όριο επάρκειας, το οποίο σημαίνει ότι πλέον δεν είναι βιώσιμο από αυτή την έννοια το εξωτερικό σύστημα. Άρα βλέπουμε ότι βιωσιμότητα και επάρκεια είναι οι δύο ψωνό νομισματός. Δεν μπορούμε να τι ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι επαρκές, ότι είναι μάλλον ε, βιώσιμο ένα σύστημα χωρίς να είναι επαρκές. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να εξετάσουμε και με ρεαλιστικό βέβαια βλέμμα τι ε, συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι αηφόρα, τα οποία ναι, μπορεί με να θεωρηθούν αηφόρα βραχυπρόθεσμα γιατί έχουν πολύ χαμηλέ παροχέ για το σταξιούχο, αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι ούτε αυτά αηφόρα. Βιώσιμα δηλαδή. Και άρα χρειαζόμαστε εξ αρχή ε, βιώσιμα συστήματα τα οποία μας προσφέρουν ε, σε βάθος χρόνου, όπως θα λέγαμε, επαρκή σύνταξη για τους πολίτες. Και Τώρα θα ήθελα να περάσω, μου επιτρέπετε, στα 14 ερωτήματα που έχουμε συμπεριλάβει στην Πράσινη Βίβλο. Μια τελευταία φορά τις κυβερνήσεις ε, για μια ευρωπαϊκή πολιτική συντάξεων. Θα επανέλθω στο τέλος. Οι άλλες 13 ερωτήσεις λοιπόν μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις κυρίως τομείς. Τα πρώτα τέσσερα ερωτήματα έχουν μάλλον χαρακτήρα στρατηγικό για την ε, συνταξιδοτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα εδώ να κατέσω σαφές ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα θέματα της ταξιδιωτικής πολιτικής. Πολλά ανήκουν μόνο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως εμείς με την στρατηγική αυτή, για τα ερωτήματα για τη στρατηγική, συζητούμε όχι μόνο τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε τι θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λιέγη, το σχετικό συμβούλιο και ένα μόνο παράδειγμα ε, το σχετικό με την πρώτη ερώτηση, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, επάρκεια, όπου έγιναν πολλές συζητήσει για το αν θα πρέπει να επιβληθεί παραδείγματι μια σειρά ή να εισαχθεί μια σειρά αρχών, προδιαγραφών του τι σημαίνει επαρκή σύνταξη τι θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές για συντάξεις στην Ευρώπη. Ναι, περίπλοκο βέβαια το θέμα, γιατί τα σταξιδιωτικά συστήματα διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αλλά αυτό ήταν για να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο του ε, διτού χαρακτήρα των ερωτημάτων που θέτουμε. Δηλαδή και γραμμή πολιτικής πώ θέλουμε να προχωρήσει η πολιτική μα, αλλά και σε τι μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την ε, βιωσιμότητα κατά τον ίδιο τρόπο. Η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με την αντιστάθμιση του χρόνου που μπορεί να περνάει κανεί στον χώρο εργαζόμενο, δηλαδή ε, και στη συνέχεια ω συνταξιούχο στο μέλλον η άλλη έχει να κάνει με ε, μηχανισμούς αυτόματους ή ημιαυτόματους προσαρμογής, αλλαγές ε, στην ηλικία της ταξιοδότησης. Με βασικό ερώτημα πάλι τι ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραματίσει στην υπόθεση αυτή. Και η τέταρτη γενική ερώτηση έχει να κάνει με τον ε, συσχετισμό με την απασχόληση, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει γνώση και γεγονότο ότι είναι πολύ σημαντική βέβαια η μεταρρύθμιση και τη εργατική πολιτική και τη ταξιδιωτική πολιτική. Δίνει δηλαδή καλά μηνύματα, μπορεί να δώσει σημαντικά μηνύματα στην ταξιδιωτική πολιτική και στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Αλλά μόνη τη η ταξιδιωτική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από μια κατάλληλη πολιτική για την απασχόληση και εδώ ακριβώς έχουν τη θέση του διάφορα ζητήματα σχετικά με την ποιοτική απασχόληση, με τις κατάλληλε συνθήκε απασχόληση με το ζήτημα των ανθρώπων που μένουν στον ενεργό βίο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κτλ. Απλώ δεν θέλω να τις τι λεπτομέρειες. Και μετά έχουμε άλλου τομεί. με τις ερωτήσεις μας, ε, παραδείγματι ζητήματα κινητικότητας, που εξετάζουμε με δύο τρόπους, είτε ως κινητικότητα των ε, συνταξιδοτικών συστημάτων, συνταξιδοτικών ταμείων καλύτερα, δηλαδή ένας τρόπος να ενισχύσουμε την κινητικότητα των πολιτών θα ήταν να έχουμε ε, συνταξιδοτικά συστήματα τα οποία θα ξεπερνούν τα πλαόρια των ε, κρατών μελών και αντίστοιχη νομοθεσία βέβαια και δεύτερο, που ίσως γνωρίζει καλύτερα η Επιτροπή σας, είναι το ζήτημα της ε, μεταφοράς εξωτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όπως μπορεί να αλλάζει ε, κατοικία ο ε, συνταξιούχος ή ο δικαιούχος να μπορεί να μεταφέρει και τα εξωτικά του δικαιώματα. η λεγόμενη οδηγία περί μεταφοράς ε, που έχει μείνει εκκρεμής ακόμη στο Συμβούλιο και που ξέρω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο γενικά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει αρκετά στο Συμβούλιο. Θέτουμε λοιπόν τα σχετικά ερωτήματα εδώ. Μετά έχουμε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των συντάξεων. που επίσης χαρακτηρίζεται πιστεύω από την εμπειρία που έχουμε λόγω και της οικονομικής κρίσης χωρίς ε, να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες θα αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία μόνο έχουμε διάφορα συστήματα ως προς τη χρηματοδότηση, άλλα ρυθμιζόμενα, άλλα μη και ρωτούμε εάν θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο συστηματική ρύθμιση των διατάξεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εν προκειμένου στην πράσινη βίβλο υπενθυμίζονται οι δεσμεύσεις του G20. Επίσης, Εάν κοιτάξουμε όλα αυτά από, το, από την οπτική γωνία του κοινού, θα έλεγα, πολίτη, του απλού ανθρώπου, που δεν αντιλαμβάνεται ίσως ε, όλες τις πτυχές ε, των ε, συστημάτων που, από τα οποία έχει να επιλέξει, στο και αν κάποιος είναι οικονομολόγος μπορεί να μην γνωρίζει κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια των συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να υπάρχει μια δυνατότητα για εξισορρόπηση των κινδύνων του της παροχής των εισφορών της ε, βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά εάν αυτά τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκά ή δυνάμει ευρωπαϊκά. Και εν των συζητήσεων και του διαλόγου που αναπτύχθηκαν ε, λόγω και της οικονομικής κρίσης. Επίσης, τα λεγόμενα ανταποδοτικά συστήματα όπου το κίνδυνο ουσιαστικά επι, ε, επομίζεται το ίδιο το άτομο, ο ίδιος ασφαλισμένος, όπου πάλι είναι πολύ πιο σημαντικό το ζήτημα της ε, ε των συστημάτων. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στο σύστημα των εισφορών όπου τον κίνδυνο έχει ο ίδιος, ε, με τον, κίνδυνο επομένως το ίδιο ο εργοδότης. Εδώ λοιπόν ίσως θα πρέπει να δούμε ε, διαφορετικές λύσεις και κυρίως κανόνες φερεγγιότητας για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Έχει ανοίξει το πεδίο για διάλογο. Περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Ξέρω ότι είναι πολλά θέματα. Ε, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης και το πρόβλημα της, όχι μόνο της φορογκαιότητας, αλλά πέραν αυτής της πάυσης πληρωμών ή και της πτώχευσης, που βέβαια δεν συμβαίνει καθημερινά, αλλά συμβαίνει πότε πότε και το, όταν συμβαίνει δημιουργεί πολλά προβλήματα. Θα θυμάστε ότι σε ορισμένα συνέβη αυτό το 2008-2009. Τι γίνεται λοιπόν όταν υπάρχει ε, κίνδυνος ή εμφανίζεται πάυση πληρωμών ή πτώχευση κάποιων τέτοιων ταμείων. Επίσης άλλα ζητήματα που ίσως θεωρούνται πιο πρόσφατα γιατί εμφανίστηκαν πιο πρόσφατα στον ευρύτερο διάλογο. Σχετίζονται με τον κίνδυνο που επομίζεται ο ιδιώτης, το άτομο. Την περίπτωση δηλαδή όπου υπάρχουν διαφορετικά στεξιωτικά συστήματα πάλι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή ο, ο ασφαλισμένος έχει μπροστά του διαφορετικά συνταξιδοτικά συστήματα που όλα όμως του ε, μεταθέτουν τον, κίνδυνο, τον κίνδυνο. Δεν ε, ανήκει ο κίνδυνος στον εργοδότη, αλλά μόνο στον ε, ασφαλισμένο. Και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια κάποια ασφάλεια. Ναι, κάποιο μου λέει εδώ ότι δεν υπάρχει σε όλε τι χώρε αυτό το πράγμα. Όντω, αλλά σε κάποιε χώρε μπορεί να συμβαίνει. Και επίση το υποβόσκουν εδώ ερώτημα που δεν αναφέρεται ίσως ρητά στην πράσινη βίβλο, αλλά πάντως υπάρχει. Τι είναι το τι σημαίνει συνταξιωτικό σύστημα. Δηλαδή, συμφωνούμε ότι οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύνταξη και αντίστοιχα να συνοδεύεται από τις ε, φορολογικές ρυθμίσεις ή τις ενισχύσεις που μπορεί να προσφέρει το κράτος. Και τι σημαίνει σύνταξη. Σημαίνει κάποια πρόσοδο μέχρι τέλους ε, του βίου, από την ώρα της σύνταξης και μέχρι το θάνατο υπάρχουν τακτικές πληρωμές. Αυτό είναι. Υπάρχουν διάφορα συστήματα όμως που μπορεί να ονομάζονται ακόμα σύνταξη, χωρίς όμως να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα ενός τακτικού, δηλαδή ενός τακτικός καταβαλλομένου ποσού μέχρι το τέλος του βίου. Αυτά πρέπει να τα ξαναεξετάσουμε. Επίση, το, ζήτημα, το ζήτημα τη διαχείριση στο μέλλον των συνταξιδοτικών συστημάτων. Που έχουν σχολιάσει και κάποιοι δημοσιογράφοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο για αυτή τη λεγόμενη ολιστική προσέγγιση στα στρατιωτικά συστήματα που θα επιτρέψει σε όλους τους παράγοντες να συζητήσουν ανοιχτά και να καταλήξουν βεβαίως το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τα σημαντικά θεσμικά όργανα δηλαδή που διαδραματίζουν ρόλο πρωταρχικό στην υπόθεση αυτή, αλλά και η κοινωνική και η οικονομική εταίρεια, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, η ενώση των καταναλωτών κτλ. Σταματώ εδώ λέγοντας ότι οι διαβουλεύσεις κλείνουν στις 15 Δεκεμβρίου Ξέρω ότι για ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, αλλά μικρό για το κοινοβούλιο και τη δυνατότητά σας να διατυπώσετε γνωμοδότηση. Ελπίζουμε όμως ότι θα μπορέσουμε να έχουμε χωρίς μεγάλη καθυστέρηση το, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου ή αμέσως μετά τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή είναι, σε, είναι διατεθειμένη να αντιδράσει, όπως είπα και ο Πρόεδρος μέσα στο πρόγραμμα του 2011, αλλά βέβαια ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε σε απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να έχουμε τις θέσεις σας ε, ε, εν ώψη αυτής της νέας πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού δώσουμε το λόγο στον δεύτερο προσκεκλημένο μας. Θα ήθελα και εγώ να πω κάποια λόγια ή μάλλον να δώσω πρώτα το λόγο κατευθείαν στον εκπρόσωπο του ΟΣΑ, τον κύριο Whitehouse, ο οποίος θα μπορέσει να απαντήσει και στα όσα είπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναφερθεί επίσης και στις ε, έρευνες, μελέτες, ε, συγκεκριμένε αναλύσεις που έχει κάνει ο ΟΣΑ όσον αφορά το ζήτημα αυτό των ε, συντάξεων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η γενική συζήτηση. Κύριε Whitehouse, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα εγώ να ορίσω τον ε, όρο ολιστικός, αλλά όπως είπε και ο κύριος Φίσερ, περιέγραψε πολύ καλά πως ε, τα συνταξιδοτικά συστήματα αντιμετωπίζονται από διαφορετικές ε, υπηρεσίες στις Βρυξέλλες. Πάντως, έχω πάει σε πολλές ε, χώρες και νομίζω ότι αυτό κάνουν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Στον ΩΣΑ υπάρχει μια ομάδα εργασία για τις ε, ιδιωτικές συντάξεις, αλλά και μια άλλη μονάδα για την κοινωνική πολιτική που καλύπτει και αυτή η μονάδα το ζήτημα των συντάξεων. Είναι σημαντικό λοιπόν, πιστεύω και εγώ, να υπάρχει όντω ένα μηχανισμό προκειμένου να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, καθότι τα αξιωτικά συστήματα τόσο διανεμητικά όσο και κεφαλοποιητικά γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και βέβαια έχουν ως στόχο να παρέχουν ένα επαρκές εισόδημα σε προχωρημένη πια ηλικία. Θα ήθελα να πω ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ενδιαφέρον και βασίζεται στις τρεις αυτές βασικές αρχές επάρκεια, βιωσιμότητα και ασφάλεια. Ο κύριος Φίσερ αναφέρθηκε στο πώς επάρκεια και βιωσιμότητα είναι διόψεις του ίδιου νομίσματος και όντως αν οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλές και όταν υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια, τότε κοινωνικά από κοινωνική πλευράς το εξωτερικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και αν οι συντάξει είναι πάρα πολύ υψηλέ όμω και κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, τότε αργά ή γρήγορα θα υπάρξει κάποια αντίδραση, θα πρέπει να επιβληθεί κάποια μεταρρύθμιση και αν αργήσει η μεταρρύθμιση, τότε θα υπάρχουν δυσμενείς αποφάσεις και αυτές θα πειράσουν επίσης και την συμπεριφορά των ίδιων των ανθρώπων όσον αφορά τις αποφάσεις αποταμίευσης για παράδειγμα που θα λάβουν. Πάντως, ε, όντως, υπάρχει μία αλληλεξάρτηση μεταξύ επάρκειας και βιωσιμότητας. Θα πρέπει κανείς, εφόσον επενδύει πολύ σε γενόδορες συνταξιωτικές παροχές, αυτές οι παροχές να είναι και βιώσιμες. 14 είναι οι ερωτήσεις του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θα τις αναλύσω όλες. Πάντως η πρώτη ερώτηση πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει να κάνει με τον καλύτερο ορισμό τη βιωσιμότητα ή αν πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει καλύτερα τη βιωσιμότητα. Η δική μου απάντηση είναι ναι. Με τον όρο επάρκεια ε, εννοούμε πολύ διαφορετικά πράγματα πολλές φορές. Πολλοί θεωρούν ότι μέσω της ε, επάρκεια εννοούμε απλώ ότι αν έχουμε μηδενική φτώχεια τα αστυνομικά συστήματα θα είναι επαρκή. Από την άλλη υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ποσοστό αναπλήρωση, δηλαδή ότι καθένα θα πρέπει να έχει ένα εισόδημα και στη συνέχεια μία σύνταξη η οποία ανταποκρίνεται στον μισθό του. Ορισμένοι λένε ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι 60%. Ο Διεθνή οργανισμό εργασία λέει ότι το μήνυμο ποσοστό τη σύνταξη θα πρέπει να είναι το 40% του τελευταίου μισθού το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την ε, μεταρρύθμιση του δικού του εξωτικού συστήματος αποφάσισε να απευθυνθεί στους ίδιους τους ανθρώπους και είδανε ότι ε, οι πολίτες με μεσαία εισοδήματα θέλανε κατά τη διάρκεια της ταξής να έχουν τα ίδια χρήματα που είχαν και όταν εργάζονταν. Αυτοί με το χαμηλό εισόδημα θέλανε πάνω από το 100% του εισοδήματος που είχαν όταν εργάζονταν, 140% συγκεκριμένα ζήτησαν, ενώ οι πλούσιοι τελικά είπαν ότι μπορούμε να ζήσουμε και με λιγότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της ε, σύνταξής μας. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα της επάρκειας θα πρέπει να καλύπτει και άλλα πράγματα, να μην αναφέρεται απλώς στην εξάλληψη της φτώχειας ή στη μη ύπαρξη ένδυας, προκειμένου να μην επηρεάζει αυτή της ε, συντάξης, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται και σε ένα καλύτερο συντονισμό του όλου συστήματος. Εμείς έχουμε κατατάξει τις χώρες σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες όσον αφορά τις ε, παροχές που δίνονται προς τους συνταξιούχους και σε ορισμένες χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Πορτογαλία για παράδειγμα, αλλά έχουμε και την Ιαπωνία και την Τουρκία, έχουμε περικοπές που γίνονται σε διάφορους τομείς. Το ίδιο ποσοστό δηλαδή περικοπής εφαρμόστηκε σε όλες τις κατηγορίες πολιτών, είτε ήταν ε, χαμηλόμισθοι είτε είχαν υψηλούς μισθούς. Υπήρχαν άλλες χώρες οι οποίε προσπαθούσαν να εξορροπήσουν καλύτερα τις, τα εισοδήματα κατά τη διάρκεια του σύνταξης και τα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ενεργούς ζωής. Σε αυτές τις χώρες έχουμε την Ουγγαρία και την Ιταλία για παράδειγμα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ω βάση μια ευρύτερη αντιμετώπιση της έννοια τη επάρκεια. Και έχουμε και δύο ακόμα κατηγορίες μεταρρυθμίσεων, όπου έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες προχώρησαν σε περικοπές αλλά προσπάθησαν να προστατέψουν τους χαμηλόμισθους. Για παράδειγμα η Φιλανδία, η Σουηδία, η Γαλλία ανήκουν στις χώρες αυτές. Και έχουμε και κάποιες χώρες οι οποίες αύξησαν τις παροχές, τις συνταξιδοτικές αλλά δώσαν κυρίως τις υψηλότερες αυτές παροχές στους χαμηλόμισθους. Έχουμε για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και άλλες χώρες στην κατηγορία αυτή. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα χώρες οι οποίες προσπάθησαν να αποφύγουν την εξορόπηση αυτή επάρκειας και βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας περισσότερο διανεμητικά στα συστήματα και προσπαθώντας να υποστηρίξουν τους χαμηλόμισθους. Αν δούμε τώρα το σύνολο των κρατών του ΩΣΑ, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την Ολλανδία και την Τσεχία που έχουν την τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας κατά τη διάρκεια της σύνταξης με ένα ποσοστό περίπου 4%, αλλά έχουμε και πολλές χώρες που έχουν χαμηλές δεξιωτικές δαπάνες. Στη Τσεχία είναι 7% του εθνικού εισοδήματος, ενώ σε άλλες χώρες έχουμε το 4-5% μόνο, σε σύγκριση με το 9% που έχουμε σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί λοιπόν κανείς να συνδυάσει τις χαμηλές ταξιωτικές παροχές με ένα βιώσιμο και παρκές στεξιωτικό σύστημα. Επίσης, στην προσπάθεια του ορισμού του όρου επάρκεια, είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα και τον όρο βιωσιμότητα, γιατί ο όρος βιωσιμότητα μπορεί να έχει διαφορετικές ε, έννοιες. Υπάρχουν ορισμένε χώρε που μπορούν να επιλέξουν να δίνουν υψηλότερε συντάξει και επομένω να ζητήσουν και τι υψηλότερε εισφορέ που χρειάζεται για ένα τέτοιο, σύστημα. Άλλε χώρε μπορούν να επιλέξουν το αντίθετο. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα επιλογών, αν θέλετε. Αλλά όπω είπε και ο κύριο Φίσερ στην παρουσίασή του, οι περικοπές στις μελλοντικέ παροχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας και το ζήτημα της ε, επάρκειας είναι ένα ζήτημα το οποίο θα επαναπροκύψει. Αν δούμε τώρα τα δεδομένα πριν από τρία, ε, 30 χρόνια, με συγχωρείτε, τα ποσοστά ένδυας ήταν ιδιαίτερα υψηλά και νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της κοινωνικής πολιτικής των τελευταίων 50 χρόνων είναι η μείωση της ε, φτώχειας των ποσοστών ένδυας στους ε, συνταξιούχους. Είναι σημαντικό βέβαια να δούμε τι εξέλιξη υπάρχει σε αυτή τη... Το έγγραφο επίσης αναφέρεται στην ηλικία συνταξιοδότησης και νομίζω ότι ε, η αύξηση του ορίου εξοδότησης είναι ο λιγότερο επιζήμιο ε, τρόπο για να μεταρρυθμίσει κανεί τα συντηρητικά συστήματα. Λιγότερο επιζήμιο, αν θέλετε, ή επώδυνο από ότι οι περικοπέ, η μείωση των συντάξεων. Από τη δεκαετία του 60 μέχρι την, το τέλος της δεκαετίας του 1990 ε, το σεξουαλικό έτος για τους άντρες ήταν 62,5 χαμηλότερο για τις γυναίκες ηλικία αυτή έχει αυξηθεί έκτοτε, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές χώρες οι οποίες ε, ε, λάβαν τις απαραίτητες νομοθετικές αποφάσεις προκειμένου να αυξηθεί το ε, έτος συνταξιοδότηση. Ο μέσος όρος θα είναι 64 για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050. Έχουν εφαρμοστεί ήδη σε ορισμένε χώρε αυξήσει τη της ηλικία αλλά και αυτέ πάλι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την αύξηση του προσδοκίμου ζωής. Μέχρι το 2050 οι άνδρες θα προσθέσουν κόμμα έτη στα αξιοδότηση στη ζωή τους, οι γυναίκες 1,5 έτος. Οι αυξήσεις σε χώρες όπως η Τσεχία και η Δανία Μάλλον στι χώρε αυτές έχουν ήδη γίνει μεταρρυθμίσεις. Σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο οι μεταρρυθμίσεις έχουν περισσότερο ως χρονικό ορίζοντα το 2050 ή το 2040. Και υπάρχουν ακόμα 11 χώρε που δεν έχουν νομοθετήσει για την ηλικία εξοδότηση για τι γυναίκες, δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή σε μια μεταρρύθμιση. Ορισμένες χώρες προσπάθησαν να συνδυάσουν άμεσα τις παροχές και την ηλικία εξοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, με την αύξηση προσδοκίμου ζωής, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, ανάμεσα στις χώρες αυτές και η Γερμανία, Ουγγαρία, Σουηδία και η Σλοβακία έχουν ε, νομοθετήσει ακολουθώντας αυτό το δρόμο. Για να καταλήξουμε τώρα, να, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ομάδα του κυρίου Φίσερ για, το πολύ ενδιαφέρον αυτό έγγραφο. Όντως θα με ενδιαφέρει και εμένα να δω πώς ε, ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της ε, διαβούλευσης και θα ήθελα πολύ να δω τι, πώς θα δημορφωθεί το έγγραφο αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτές τις δύο παρουσιάσεις. Πολύ πλήρης. Θα περάσουμε στη συζήτηση. Πρώτα, κυρία εισηγήτρια, κυρία Όμεν Ρόιτεν, παρόλο που στην ημερήσια δεν είχε ακριβώς με αυτή τη μορφή το σημείο αυτό, επειδή δεν αριθμίσαμε ακόμα το θέμα της αρμοδιότητας με την Οικονομική Επιτροπή. Δεν το ανακοινώνουμε λοιπόν επίσημα. Αλλά υπενθυμίζω όπως και η Κομισιόν που ασχολείται με αυτό το φάκελο. Ελπίζω και οι υπόλοιποι να κινητοποιηθούν ώστε να γίνει αυτό που θέλουμε. Κυρία Ομετρόιτη και μετά κυρία Κάστεξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, πολύ ωραία. Αν εσείς θα μπορούσατε να ζητήσετε αυτό το έγγραφο για μας, θα ήταν πολύ καλό επειδή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε την Γενική Υπόθεση Κοινωνικών Υποθέσεων. Νομίζω ότι ε, εσεί έχετε αρκετή δύναμη να πετύχετε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση και η Οικονομική Επιτροπή να συντάξει αυτή με τη σειρά τη μια γνωμοδότηση. Είναι βέβαιο ότι θα συνεργαζόμασταν αν κάποιο από αυτήν την Επιτροπή την Οικονομική θέλει να γράψει μια γνωμοδότηση. Δεύτερη παρατήρηση. Όλο αυτό το θέμα των συντάξεων είναι πολύ ευρύ. Είναι πολύ μεγάλο. Θα πρέπει λοιπόν να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε καλά μεταξύ μας. Επειδή υπάρχουν τεράστιες διαφορές αναχώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα καλέσω όλους όσους έχουν κάτι να πούνε σε αυτό το θέμα ή κάποια συμβολή να συνεισφέρουν να το κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο ως Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να χαθούμε σε ένα είδος μπερδεμένων ιδεών και συνοθηλεύματος που δεν μας αφήνει δηλαδή να έχουμε μια ομοιογενή και ξεκάθαρη θέση και άποψη εδώ στην ομάδα μας. Τώρα, μιλώντας βεβαίως για το θέμα της δαξιοδότησης και των συνταξιοδοτικών ταμείων, με όλα αυτά τα θέματα της κρίσης και τα λοιπά, διερωτάται κανείς ποιο είναι το κοινωνικό υπόβαθρο εδώ. Εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο οι συντάξει θα πρέπει να είναι αξιοπρεπεί και να τουλάχιστον να συντίζουν τον κόσμο ώστε να μην πεθαίνει τη πείνα. Θα πρέπει εκτό από αυτό να, να πούμε ότι είναι ένα κεντρικό σημείο τη κοινωνικής μας ζωής. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ, όπου πολύ σύντομα για κάθε εργαζόμενο θα λείπουν άλλοι δύο εργαζόμενοι, τότε οι ελλείψεις που θα υπάρχουν είναι τεράστιες. Όσοι λοιπόν βρίσκονται σε μια ενεργό εργατική ζωή θα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί με τη σειρά του ότι δεν πιούν μόνο για του εαυτού του αλλά και για τι επόμενε γενιέ. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξουν τα συμφέροντά του. Και αυτό λόγω και τη γύραση τη κοινωνία. Οπότε πώ θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μελλοντικά συστήματα συνταξιδοτικά για το μέλλον που να είναι πιστευτά και εφαρμόσιμα. Δεύτερη ερώτηση για τον προπολογισμό. Επισερχόμενοι και σε κάποια θέματα νομισματικά. Πρώτον, θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο η Ευρώπη έχει αρμοδιότητα για το θέμα των συντάξεων και εγώ νομίζω ότι κάλλιστα την έχει. Επειδή η κινητικότητα μεταξύ των Ευρωπαίων αυξάνεται συνεχώς, αυτό σημαίνει ότι όσοι πάνε να εργαστούν σε κάποια χώρα ή να σπουδάσουν θα μπορούσαν να έχουν στη διάθεσή τους όχι μόνο μια κρατική εργασία, αλλά θα πρέπει να έχουν καταβάλει όλες τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις ώστε να μην αποτρέπονται οι εργαζομένοι από το να κινητοποιηθούν. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με την ε, κινητικότητα των πολιτών, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου το ότι ό,τι έχει βγάλει κανείς αφορά αυτό που γίνεται στις διάφορες χώρες μέλη. Αλλά ήδη υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να ιδιοποιηθεί τέλο πάντων ή να αφαιρέσει ένα σημαντικό κομμάτι των μισθών. Οπότε θέλω να πω ότι αυτές οι ελάχιστες περιγραφές για την κινητικότητα θα πρέπει να μην είναι περιοριστικέ. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία ζουν σε μια χώρα και εργάζονται σε μια άλλη. Αυτά είναι θέματα κοινωνικά. Είναι και χρηματοοικονομικά. Βεβαίω, σαφέστατα, επειδή κινητοποιείται και αρκετό χρήμα ή διακινείται χρήμα. Οτιδήποτε όμως χρηματοδοτείται από το σύστημα συνταξιδότησης το κάνει να διατρέχει τον κίνδυνο ένα κίνδυνο που αφορά ας πούμε θέματα νομισματικά όταν καταβάλλεται ένα μισθό σε, σε διαφορετικό νόμισμα από ό,τι θα έπρεπε τι έγινε α πούμε στην Ελλάδα κοιτάξτε τι έγινε με τι ελληνικέ ε, συντάξει στην Ελλάδα όλα αυτά είχαν σημαντικά σημαντική απήχηση και επιπτώσει. θέλω να πω δηλαδή ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα νέο σύστημα καταβολή των συντάξεων θα πρέπει μόνο να μελετήσουμε το πώ θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε καλύτερα το σύστημα το συνταξιοδοτικό και το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε όταν μιλάμε ας πούμε για μια σύνταξη η οποία προέρχεται από ένα αργοδότη κυβερνητικό ή κρατικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αρχή η οποία θα πρέπει να ελέγχει ακριβώς τις συντάξεις αυτές. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε μια ευρωπαϊκή ή πανευρωπαϊκή οπτική για το θέμα των συντάξεων. Δεύτερον, θα θέλαμε να δοθεί αυτό σε εμά ως Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Είπε το Ολλανδικό Κοινοβούλιο πρόσφατα ότι το θέμα των συντάξεων είναι εθνικό τελεία και παύλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε κάποιες εθνικές απόψεις, αλλά δεν νομίζω να είναι εθνικό προνόμιο αυτό το θέμα μόνο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να δώσουμε μάχη ακριβώς για να περάσει και η, δική μας η δικαιοδοσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καστέξ και μετά η κυρία Τωρινέν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω και εγώ η Επιτροπή Απασχόλησης να, να είναι η κατουσία αρμόδια για την γραμμοδότηση αυτή, επειδή νομίζω ότι έχουμε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση για το θέμα των συντάξεων και όχι μόνο λογιστική, όπως ενδεχομένω έχει η Οικονομική Επιτροπή. Επειδή θεωρώ ότι ο περιορισμός της προσέγγισης που προτείνουμε εμείς προς την Κομισιόν αφορά ακριβώς το ζήτημα αυτό από μια στατιστική και οικονομική ή νομισματική σκοπιά. Δηλαδή η Κομισιόν παρουσιάζει κάποιες μαθηματικές προεκβολές σαν να ήταν ε, προγνώσεις. Το να πούμε σήμερα λοιπόν ποιο θα είναι το ποσοστό εξάρτησης μεταξύ ενεργών και ανενεργών το 2060 αφορά νομίζω μία προβολή τελείως ανώφελη. Επειδή το 2060 αυτοί που θα είναι ο ενεργός πληθυσμός δεν έχουν γεννήθει ακόμα. Οπότε τα επόμενα χρόνια λοιπόν θα δούμε πώς θα έχει εξελιχθεί και το το γεννήσεων. Προς το παρόν δεν μειώνεται στις διάφορες χώρες μέλη. Πάντως αυτή τη στιγμή όταν έχουμε μείωση, δεν μπορούμε να πούμε κατά πόσο έχουμε μία μείωση ουσίας ή απλά και μόνο μία καθυστέρηση στην γέννηση του πρώτου παιδιού όπως παρατηρούμε όπω παρατηρούμε σε διάφορε χώρε όπω η Γαλλία. οπως παρατηρουμε σε διαφορε χωρε οπως η γαλλια οποτε το να βασίσουμε ένα ολόκληρο σύστημα και ολόκληρα συμπεράσματα σε αυτό το είδος ε, προβολών ε, θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της εξάρτησης αλλά και για το θέμα της ε, απασχόλησης, δηλαδή την ενεργό ζωή. Νομίζω ότι ε, δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοια ποσοστά ανεργίας όπως αυτά που έχουμε σήμερα. Και αν δούμε αυτά τα ποσοστά, τότε θα κατανοήσουμε ότι για να αυξήσουμε τον ενεργό πληθυσμό έχουμε κάποια περιθώρια αύξησης της απασχόλησης για τους νέους, για τους ε, ηλικιωμένους, για τις γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε και ένα σενάριο σύνταξης με προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνουν και την πλήρη απασχόληση. Νομίζω ότι η καθαρολογιστική προσέγγιση βασιζόμενη μόνο στους ε, μισθωτούς απομακρύνει το ενδεχόμενο να, χρηματοδοτούνται οι συντάξεις από άλλες πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή πέραν των κοινωνικών εισφορών που θα βασίζονται τέλο πάντων στις εισφορές του μισθού. Μέχρι το 2060 θα μπορούσαμε να προβλέψουμε την ύπαρξη ενός μιας προσθέμενης αξίας στον πλούτο που δημιουργείται και αυτό δεν το αναφέρει το, πράσινο βιβλίο. Τώρα, τούτου λεχθέντος, νομίζω ότι μία από τις κυριότερες επικρίσεις που θα έβλεπα εδώ είναι καταρχήν το ότι ακολουθούμε μια προσέγγιση που δεν είναι ίσως η κατάλληλη όσον αφορά την σταξιδότηση και το προσδόκιμο ζωής. Γιατί βεβαίως ε, έχουμε διάφορες εκθέσεις που λένε θα πρέπει να θεσπίσουμε τον κύκλο της ε, ενεργού ζωής. Εδώ όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ηλικία σταξιδότηση ακριβώς για να προσεγγίσουμε το θέμα της σύνταξης γενικότερα και το θέμα των εισοδημάτων από σύνταξη σε σχέση με μια γενικότερη προσέγγιση της, ενε, της ε, ενεργητικής ζωής όσον αφορά τη διάρκεια της εργασίας και τα λοιπά. Τότε λοιπόν από την Κομισιόν θα είχαμε κάποιες χρήσιμες ενδείξεις Θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν κάποιες ενδείξεις για την ενεργό ζωή, για το flex security, για το πώς θα μπορούσαν να είναι βιώσιμα αυτά τα συστήματα, τα συνταξιδοτικά, σε μια περίοδο όπου η ενεργός ζωή εξελίσσεται με κάποιες μετεξελίξεις ή εναλλαγές, ενεργό ζωή, κατάρτιση, ανεργία κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε πώ ακριβώς αυτοί που εναλλάσσονται στα διάφορα ενεργητικά στάδια της ε, επαγγελματική του ζωής, πώ θα μπορούσαν λοιπόν να χρηματοδοτήσουν ή να κάνουν ό,τι χρειάζεται τέλο πάντων ώστε να έχουν στη διάθεσή τους μια αξιοπρεπή σύνταξη στο τέλος. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε λεπτομερέστερα το θέμα του προσδόκιμου ζωή. Αυτό είναι ένα θέμα που εμένα μου προκαλεί κάποιες ε, αμφιβολίες, κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια τακτική και αναπόφευκτη άνοδος του προσδόκιμου ζωής. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει κάπως να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής και εδώ ακριβώς θα μπορούσε να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή μιλάμε για ένα προσδόκιμο ζωής για ποιους. Αυτό το προσδόκιμο ζωής πώς ακριβώς ποικίλει σύμφωνα με την φύση της εργασίας. Ποια είδη εργασίας μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. Ποιο προσδόκιμο ζωής έχει κάποιος ο οποίος σταματάει να δουλεύει στα 60 και ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής για κάποιον ο οποίος τέλο πάντων σταματάει στα 65 ή κάποιον που σταματάει στα 67. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εργασία που γίνεται μεταξύ 57 και 67 έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στο προσδόκιμο ζωής, για το προσδόκιμο ζωής σε σχέση με εργασία η οποία γίνεται ή έχει κάποιος μεταξύ 20 και 30 ετών ηλικίας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει ακριβώς να κάνουμε λεπτομερέστερες αναλύσεις σε σχέση με αυτό το πρόβλημα ώστε να είμαστε ρεαλιστικοί στι αποφάσεις μας. Ευχαριστώ η κυρία Τρούνα και μετά ο κύριο Κοφεράτη. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον να διαβάσουμε αυτή την πράσινη βίβλα από την Κομισιόν. Πραγματικά θίγουν πολύ σημαντικά ερωτήματα και κέρια ερωτήματα για το μέλλον. Και όπως είπε και η συγγήτρια, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι όλη εδώ η προσπάθεια θα πρέπει να καθορίσει ακριβώς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το θέμα αυτό και την προσθεθήμενη αξία που θα μπορούσε να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι συντάξει, όσον αφορά επίση και την κοινοτικότητα και, το, και την ασφάλεια τη εργασία κλπ. Εδώ βεβαίω δεν θα πρέπει να καταστρέψουμε ό,τι είναι αποτελεσματικό, ό,τι λειτουργεί καλά μέχρι τώρα και να πω ότι η πράσινη βίβλο παρουσιάζει κάποια θετικά στοιχεία όσον αφορά τη βιωσιμότητα αλλά ενδεχομένω να αποφεύγει να εξετάσει καλύτερα το εργατικό περιβάλλον και την κινητικότητα και την σύνδεσή τους γιατί ακριβώς δεν έχουμε υπολογίσει τις επιπτώσεις τους στην γενικότερη οικονομία. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να το εξετάσουμε στα πλαίσια της πράσινη, πράσινης βίβλου. Δεύτερον, η ευέλικτη συνταξιοδότηση θα ήταν και αυτή κάτι το πολύ σημαντικό, επειδή κανείς θα μπορούσε να έχει δουλέψει ολόκληρη τη ζωή του και να σταματήσει τα 55 αλλά θα μπορούσε ενδεχομένω να συνεχίσει μέχρι τα 75 ε, ανάλογα με, την, ε, με του ή, ή την όρεξή του. Τώρα, η την ορεξη του τωρα η ερωτηση που έχω προς την Κομισιόν είναι η εξή. Ποιος θεωρείται θα είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ακολουθώντας την, το χρονοδιάγραμμα που θέσατε επειδή νομίζω ότι για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε περισσότερο χρόνο συνεργασίας μαζί σας πρώτον δεύτερον προς την συγκέντρια θα ήταν ενδιαφέρον νομίζω να διερευνήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα επειδή ακριβώς οι αρμοδιότητες έχουν εθνική βάση και θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια για αυτό το θέμα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια θετική ιδέα, μια καλή ιδέα. έχουμε και το πνεύμα τη συνθήκη Λισαβόνα που φέρνει το κοινοβούλιο πιο κοντά σε αυτά τα θέματα. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε βεβαίω κάλλιστα ω Επιτροπή κοινωνικών θεμάτων ώστε να δούμε καλύτερα και μελλοντικά και τα θέματα της ε, οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτ και μετά ο κύριος Σουρή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε όπως κάνει η Πράσινη Βίβλος το θέμα των συντάξεων επειδή θεωρούμε ότι αυτό αυτό το θέμα είναι από τα πιο ευαίσθητα, από τα πιο λεπτά, όχι μόνο σήμερα, αλλά και για το μέλλον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια προσέγγιση σωστή, επειδή ξεκινάμε από θέματα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους και που είναι ο καρπός της ιστορίας και δεν ταυτίζονται καθόλου. Οπότε το να προβλέψουμε κάποιες μορφές ε, παράλληλες ώστε να συνοδεύουν αυτές οι μορφές την ε, προσέγγιση την χρονική του θέματος της σύνταξης. Εντάξει, αυτό είναι απαραίτητο, αλλά αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο. Και νομίζω γι' αυτό ακριβώ το λόγο έκανε πολύ καλά η Κομισιόν να θέσει το θέμα της βιωσιμότητας με, το θέμα της επάρκειας που επανειλημμένως θεωρήθηκαν ως δύο θέματα τελείως διαφορετικά και αυτό δείξει, βεβαίω στο να υπάρχουν ε, ανισορροπίες, να υπάρχει δηλαδή έλλειψη ισορροπίας στις δημόσιε δαπάνε και που σε περαιτέρω δυσκολίε. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι στη συζήτηση θα πρέπει να εμβαθύνουμε και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι η Κομισιόν ακολουθεί τον δρόμο των πολλών ερωτήσεων με τις οποίες προσβλέπεις απαντήσεις από τους ε, συνομιλητές και θα ήθελα και εγώ να κάνω και εδώ κάποιες ε, σκέψεις. Όταν μιλάμε για απασχόληση, βέβαια θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας έναν ε, δείκτη πολύ έτσι δυναμικό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μας ανησυχεί το θέμα των συντάξεων επειδή ακριβώς στα πλαίσια μιας πολύ σημαντικής και σοβαρής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε το θέμα έχει γίνει πολύ πιο οξύ από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Από την άλλη μεριά υπάρχουν βεβαίως και τα θέματα όπως η αύξηση του προσδοκιμού ζωής που σημαίνει ότι το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στις ε, εισφορές και στην ηλικία δεξιότητες, αλλάζει συνεχώς. Αυτό ήδη θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο να επικεντρωθούμε σε κάποιες αξιολογίες οι οποίες δεν προβλέπουν ως τελική λύση κάτι το τρακόντιο. Αντίθετα θα πρέπει να εισαγάγουμε κάποια στοιχεία ευελιξίας. Όταν μιλάμε επί παραδείγματι για την βιωσιμότητα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο φαινόμενο όπως η παράνομη εργασία το οποίο αφαιρεί από τα συστήματα πρόνοιας ένα σημαντικό ποσό ή ποσοστό εισφορών. Η παράνομη εργασία έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά παρουσιάζει πάντοτε κάποια αρνητικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα εντοπίσουμε προσεκτικά. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο να επικεντρωθούμε στην αύξηση των εισφορών, κάτι το οποίο ε, απορρέει από την αύξηση της εργατικής ζωής, της ζωής δηλαδή εργασίας, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο και από την παράνομη εργασία πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις εισφορές. Όλα τα συστήματα ξεκίνησαν από την ε, διανομή και πήγαν στην κεφαλαιοποίηση. Δεν νομίζω θα έπρεπε να προβλέψουμε μία επιστροφή στα παλαιά πρότυπα. Αν όμως η κεφαλαιοποίηση αποτελέσει την βάση του επόμενου συστήματος συντάξεων οι συνταξιδότηση, τότε θα πρέπει να έχουμε επίγνωση από τώρα, από τώρα ότι η δημόσια πρόνοια δεν θα είναι ποτέ επαρκής για να απαντήσει σωστά στις ανάγκες ή στις απαιτήσεις επάρκειας που υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τρεις πυλώνες. Ο δημόσιος πυλώνας που θα βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση. Ένας πρώτος πυλώνας ιδιωτικός, ο οποίος θα απορρέει από την αποταμίευση, δηλαδή από το ποσό εκείνο που οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα μπορούσαν να το προορίσουν στην πρόνοια. Και θα χρειαστεί επίσης και ένα σύστημα κινήτρων σε ένα ενδεχόμενο τρίτο πόλο, μάλλον πυλώνα, συγγνώμη, απαραίτητο μάλλον, που είναι η ιδιωτική αποταμίευση. Δηλαδή σε περίπτωση όπου κάποιος θα ήθελε να έχει περισσότερη εξασφάλιση σε σχέση με το μέλλον, τότε μια φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με αυτό το τρίτο πυλώνα θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη και να είναι διαθέσιμη ως εργαλείο στις κυβερνήσεις. Μια τελευταία σκέψη για την κινητικότητα. Επειδή η κινητικότητα αναφέρθηκε επανειλημμένω, η κινητικότητα όμω για την οποία θα πρέπει να μιλάμε δεν είναι αυτή που είχαμε πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ δεν αφορά την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Επειδή βρισκόμαστε ενώπιον ενό αυξανόμενου φαινομένου κινητικότητα ατόμων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Δηλαδή εργάζονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά επαναπατρίζονται με τον στόχο βέβαια να πάρουν μαζί τους και τα ποσά τα οποία κατέβαλα και το οποίο θα ήθελα να μεταφέρουν στο δικό του σύστημα, στη χώρα του προέλευση. δηλαδή. Αυτό όμω θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. γιατί αν ανατραπεί η δημογραφική τάση στην Ευρώπη, τότε τα αποτελέσματα θα δούμε σε 20 και 30 χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ευρωπαίοι θα θέλουν να έχουν περισσότερα παιδιά από ό,τι είχαν τα τελευταία χρόνια. Αν όμω αυτό συμβεί, τότε τα θετικά αποτελέσματα είναι πολύ μακρινά. Οπότε εμεί θα πρέπει να έχουμε για πολλές δεκαετίες λύσει το δημογραφικό πρόβλημα με την σημαντική συμβολή ατόμων που γεννήθηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου και υπάρχουν να δουλέψουν εδώ και τα οποία δεν επέλεξαν να μείνουν εδώ για πάντα. Πολλά από αυτά τα άτομα θα, θα ήθελαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Οπότε η κινητικότητα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προλαμβάνει αυτή, ακριβώ αυτή την πιο, πολύ πιο ευρεία εξαίρεση από ό,τι, από είχε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σωρή και η κυρία Γιδασλόφσκα ε, στη συνέχεια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πράσινη αυτή βίβλος μας παρακινεί να αναλύσουμε περισσότερο το ζήτημα αλλά καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα αυτό από μόνο του και οι προτάσεις που γίνονται οδηγούν σε νέα ζητήματα. Η κυρία Καστέξ αναφέρθηκε σε πολύ σημαντικά ζητήματα, ότι θα πρέπει δηλαδή να δούμε περισσότερο την προσέγγιση που υιοθετεί αυτή η πράσινη βίβλος. Βασίζεται περισσότερο σε κάποια παραδοσιακά ευρωπαϊκά συστήματα και εν μέρη σε πιο μεσογειακά σε εξωτικά συστήματα. Βλέπουμε όμως ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ζήτημα το συνταξιδοτικό και όσον αφορά την βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιδοτικών συστημάτων, είτε πρόκειται για συστήματα στην Αμερική, είτε πρόκειται για τα ανάλογα συστήματα στην Ασία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τόσο το παραδοσιακό σύστημα συνεισφορών, όσο και άλλους στόχους όπως η μείωση της φτώχειας σε προχωρημένες ηλικίες. Επίσης, η χρηματοδότηση των συνταξιωτικών συστημάτων μέσω της φορολογίας και αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Σαφώς βέβαια τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με τους εργαζομένους οι οποίοι εργάζονται με νόμιμο τρόπο και αποτελούν τελικά τους βασικούς ε, πυλώνες του συστήματος. Υπάρχουν ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης. Στις χώρες αυτές δεν ξέρω αν ε, η προσέγγιση την οποία θέλουμε να υιοθετήσουμε εδώ θα μπορούσε να ισχύσει, γιατί ε, Ενδεχομένω στις χώρες αυτές να πρέπει να εξετάσουμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά παράνομη εργασία που υπάρχουν. Ας μην εξετάσουμε επίσης μόνο τις δημογραφικές τάσεις, ας λάβουμε υπόψη μα το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι στο μέλλον θα καταβάλουν πολύ χαμηλές εισφορέ στα δημόσια συστήματα αστεξοδότηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι δηλαδή όλο και περισσότερο θα μετακινούνται προ τα κεφαλοποιητικά συστήματα, προ τι ιδιωτικέ ασφάλειες. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται είναι αν υπάρχει μία μόνο προσέγγιση ή αν θα πρέπει να εξετάσουμε και εναλλακτικού τρόπους να προσεγγίσουμε το ζήτημα. Αν Μάλλον η προσέγγιση αυτή που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λογιστική αυτή προσέγγιση, δεν λαμβάνει υπόψη της πολλές άλλες πτυχές του ζητήματος. Α μην ξεχνάμε ότι σε πολλέ χώρε, όπω για παράδειγμα στη Γαλλία και πρόσφατα μάλιστα, είδαμε πολύ σημαντικέ διαδηλώσει, άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούσαν στην προτινόμενη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν και αυτή η κοινωνική πτυχή να ληφθεί υπόψη. Κάθε φορά προσπαθούμε να πειράξουμε το στρατιωτικό σύστημα, η κοινωνία πάντα θα αντιδρά. Χαιρετίζω λοιπόν τις παρουσιάσεις που γίνανε. Συμφωνώ με αυτό το οποίο υπόθηκε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί, να διοργανωθεί, με συγχωρείτε, μια σημαντική συνδιάσκεψη όπου θα μπορούσε να συζητηθεί και το ζήτημα αυτό, αλλά και άλλα συναφή ζητήματα όπως ε, οι κλιματικές αλλαγές και όπου θα πρέπει ουσιαστικά να συνειδητοποιήσουμε ότι τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα δεν είναι βιώσιμα. Και πάρα πολλέ φορέ βέβαια τα τα ευρωπαϊκά συστήματα, τα εθνικά μάλλον συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέχουν πολύ το ένα από το άλλο. Υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει. Επίση έχουμε 14 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο έλλειμμα και που εξετάζουν την επιρροή που έχει το δημόσιο έλλειμμα στα εξωτικά του συστήματα. και ορισμένες νέες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφεραν να προσχωρήσουν ανταποκρινόμενες σε μια συγκεκριμένη προϋπόθεση το να μεταρρυθμίσουν δηλαδή τα παραδοσιακά διανεμητικά συνταξιωτικά του συστήματα. Χρειάστηκε λοιπόν οι χώρες αυτές να προχωρήσουν σε απαραίτητε μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που δεν κάνανε ή παλιότερε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτή χώρες, οι παλαιότερες χώρες ευρωπαικη ενωση με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες αποκλήσει μέσα στην Ένωση. Η συζήτηση που ξεκίνησε είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και καταλαβαίνετε βέβαια ότι και η οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει πολύ το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα την ηλικία ταξιδότηση. Το ζήτημα αυτό δεν αναφέρθηκε ή μάλλον αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΕΛΚ, αναφέρονται στο λεγόμενο ευέλικτο όριο ταξιδότηση, ευέλικτη ηλικία εξοδότηση, όπου ο ασφαλισμένος θα μπορεί να αποφασίζει τελικά να επιθυμεί να λάβει νωρίτερα τη συνταξή του, η οποία όμως θα έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο, είναι επιθυμεί να δουλέψει περισσότερο και να λάβει τελικά μια υψηλότερη σύνταξη. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές επιλογές. Επίσης υπάρχουν κάποιες κοινωνικές πολιτικές που μπορούν να πειράσουν την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών συνταξιωτικών συστημάτων και αυτό δεν έχει αναφερθεί στην Πράσινη Βίβλο. Κατά άποψή μου λοιπόν εκκρεμούν ακόμα πολλά ερωτήματα και νέα ερωτήματα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της ε, συζήτησης. Περισσότερα δηλαδή από αυτά τα οποία έχει θέσει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά τα οποία έχει πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Η κοινωνική διαβούλευση μάλλον η διαβούλευση που προβλέπεται για αυτή την πράσινη βίβλο με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Νοεμβρίου είναι μια διαβούλευση ιδιαίτερα σύντομη. Το ΕΛΚΑ έχει πει ότι επιθυμεί να διοργανωθεί μια ακρόαση για το ζήτημα αυτό. Και αυτό που θα ήθελα εγώ να προτείνω είναι ή δυνατόν να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε το εύρος της διαβούλευσης και προκειμένου να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφώσει καλύτερα τοποθέτησή του. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιασλόβισκα και η κυρία Κρούς στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ συγκαταλέγομαι στους αισιόδοξους και φρονώ ότι τον αγώνα αυτόν της επικράτησης της διαβουλεύσης για την Πράσινη Βίβλο θα τον κερδίσει η δική μας Επιτροπή. Γιατί δεν την Πράσινη Βίβλο, και που γίνεται λόγος για γύρανση του, Ευρωπαϊκού, του πληθυσμού της Ευρώπης, δεν γίνεται αντίστοιχα και λόγος για την μείωση της γενετικότητας. Ωστόσο, θεωρώ ότι για την λειτουργία των αναδιανεμητικών ή μεικτών κυρίως ταξιδιωτικών συστημάτων έχει ουσιαδέστατη σημασία η ε, γεννητικότητα, ο δείκτης γεννητικότητας. Αλλά θα πρέπει και αυτό να συζητηθεί. Η επασχολησιμότητα τώρα. Η πράσινη βίβλος νομίζω παραβλέπει σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της ε, ανισότητας των φύλων και της ε, εξασφάλισης της ολοκλήρωσης των στεκτοτικών δικαιωμάτων για τους πολίτες και ιδίως τις γυναίκες και πολύ συχνά βλέπουμε δυστυχώς ότι οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις επειδή ε, έλαβαν την απόφαση να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν το ζήτημα πρέπει να το συζητήσουμε. Επίσης, το ζήτημα της επαρκούς σύνταξης πρέπει να μας απασχολήσει. Έχω την αίσθηση ότι γίνεται λόγος μάλλον για τις πρακτικές που έχουν επικρατήσει και όχι για τα πραγματικά δικαιώματα που θα μπορούσε κανείς να εξασφαλίσει κατά τη διάρκεια της ε, επαγγελματικής του δραστηριότητας. Και άλλο ένα ζήτημα, ίσως θα πρέπει να δεχθούμε μία μεθοδολογία ενιαία, ταυτόσιμη σε όλα τα κρατη προκειμένου να αξιολογηθούν κατά τρόπο αντικειμενικό και ουδέτερο τα σταξιοδοκτικά συστήματα σε όλα τα κρατη Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να αφορά κάθε ηλικία, ακόμη και τους νέο εισαχθέντες στον επαγγελματικό βίο. Επίσης θα πρέπει να συζητηθεί η αυστηρότητα με την οποία θα πατάσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη εκείνα τα οποία προβαίνουν σε μεταρρύθμιση των στετιωτικών του συστημάτων, ταυτόχρονα ενισχύοντας τα εθνικά τους ελλείμματα. Η μεταρρύθμιση των συνταξιδοτικών συστημάτων, δηλαδή πιστεύω, θα πρέπει να συμβάλλει αποκλειστικά και μόνο, και με αυτή την προπόθεση να γίνεται δεκτή, στον περιορισμό του εθνικού ελλείμματος δημοκρατικού ελλείμματος. Και θα πρέπει να επιβάλλονται, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό, οι σχετικέ κυρώσει. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκέρντς. Χρειάζεται, πιστεύω, να αφήσουμε ένα χρονικό περιθώριο επαρκές, ώστε να έχουμε τη γενικότερη εικόνα και της κατάστασης και των στόχων μας για να μπορούμε να αποφασίσουμε. Είναι καλές οι προτάσεις. Βέβαια πολλά πράγματα λείπουν και βλέπω ότι προσπαθούν ε, οι πάντες να διατυπώσουν ε, ε, προτάσεις και αμφιβολίες. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εκεί που με τα ε, διατηρούνται βιώσιμα τα σταξιδιωτικά συστήματα, είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν πολιτικέ αποφάσεις και είναι πολλοί εκείνοι που μας λένε δεν είναι τώρα η ώρα για κάτι τέτοιο. αξιωτικό σύστημα πρέπει να σημαίνει αξιοπιστία και σταθερότητα. Και αυτό ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ε, ε, διάθεση των ε, ασφαλισμένων να καταβάλουν τις φορές τους. Πολύ συχνά η προτίμηση εστιάζεται σε εξελίξεις σχετικές με εκούσια συστήματα ασφάλισης. Θα πρέπει λοιπόν να, δούμε μια, να, να βρούμε μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ του χρόνου απασχόλησης και της ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά και της αναλογίας ε, ενεργών και συνταξιουχών. Ταυτόχρονα διαφυλάσσοντας την συνοχή στην κοινωνία. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορους κινδύνους και όχι μόνο το ε, γύρας ως κίνδυνο ασφαλιζόμενο. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για ηλικία συνταξιοδότησης. Ίσως όμως πέραν αυτής θα πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον, ε, θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το, το σύστημα και που δεν θα είναι μόνο το πρόβλημα της υγεία, ένα πρόβλημα υγείας ενδεχομένως, αλλά και η αδυναμία να διατηρήσει κανείς μια θέση εργασίας. Και ίσως καλό θα ήταν να οργανωθεί ένα κέντρο που θα προσφέρει στον ενδιαφερόμενο πολίτη επαρκείς πληροφορίες. Απέχουμε, ξέρω, πόρο από έναν αρμονισμένο συνταξιδοτικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως να υπάρξει επαρκή επιτήρηση, παρακολούθηση και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κυρία Μάρκιν και μετά κύριο Κάσλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πολλά έχουν ήδη υποθεί από τους συναδέλφους μου. Ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα αναλάβει την κατουσία γνωμοδότηση γιατί είναι θέματα όχι μόνο οικονομικά ή απασχόληση, αλλά και κοινωνικά πάνω από όλα ζητήματα αυτά τα οποία ε, άπτονται του ταξιδιωτικού, ενός ταξιδιωτικού συστήματος. Και όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, η σύνταξη είναι σύνταξη και ω τέτοια πρέπει να εξετάζουμε. Είναι ένα περίπλοκο βέβαια θέμα ε, κοιτάμε τα ζητήματα από την οπτική βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κινητικότητα και όλα αυτά τα οποία ε, εξέθεσαν οι συνάδελφοι νωρίτερα που είναι δεδομένα, αλλά και τη μεγάλη πρόκληση ως προς την ενδεχόμενη ανατροπή μιας, της σταθερότητας της νομισματικής που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ιδιαίτερα με δεδομένες τις πρόσφατες εξελίξεις. Αλλά ιδιαίτερη σημασία ε, πρόκληση είναι η δημογραφική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει το σημαντικό ρόλο που της ανήκει στο συνταξιδοτικό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε, καινοτόμο σκέψη, καινοτόμο θεώρηση ε, βεβαίως. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι θα μπορούσαμε και εμείς ως κοινοβούλιο να εξετάσουμε τι μπορούμε να προτείνουμε σαν ιδέες, αλλά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πολίτη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Και βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον και σε φέρει το κείμενο με έκπληξη πάντως διαπιστώνω ότι για αρκετούς πολίτες και μη κυβερνητικέ οργανώσεις ενδέχεται να είναι αποτρεπτικό, διότι το να κάτσει κανείς να διαβάσει το κείμενο αυτό χωρίς να είναι ειδικό. ουσιαστικά θα τον φημώσει, δεν θα του επιτρέψει δηλαδή να εκφέρει τις θέσεις του ε, είναι πολύ περίπλοκο δηλαδή το έγγραφος για τον ε, κοινό πολίτη συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα, ένα πιο απλό δηλαδή κείμενο το οποίο θα απευθύνεται όχι μόνο στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά στον κάθε έναν που δεν είναι ειδικό, όπως εγώ. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε μία εξέλιξη κατά την οποία ή μέρημνα για τον ηλικιωμένο από άτυπη θα περάσει αποκλειστικά στο επίπεδο της επίσημης, της τυπικής, της θεσμικής δηλαδή μέρημνας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε την άτυπη μέρημνα για όσους έχουν ανάγκη μέσα στην οικογένεια ή την κοινωνία και ταυτόχρονα εκείνους οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν κάποια θυσία επαγγελματική προκειμένου να προσφέρουν αυτή τη μέρημνα, την άτυπη μέρημνα, με απώλεια ενδεχομένω μισθού ή διακοπή απασχόληση, θα πρέπει να τους ενισχύσουμε μέσα από ένα συνταξιδοτικό σύστημα ικανοποιητικό. Και πιστεύω ότι ο συνάδελφο από τον ΟΣΑ ε, ξέφρασε την πιο σημαντική παρατήρηση ως προς τα αναδιανεμητικά στα εξωτικά συστήματα. Εδώ νομίζω θα πρέπει να εστιαστεί η συζήτηση και πολύ, με πολύ μεγάλη αδημονία περιμένω την ώρα να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες των θεμάτων αυτών. Επίσης η Επιτροπή μίλησε για την υλοποίηση της οδηγίας περί αφαιρεγγιότητας και δεν θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν εξελίξεις ε, συγκεκριμένες στις οποίες θα μπορούσε η Επιτροπή μας να εντυπώσει προτάσεις. Ο κύριος Σωρή μίλησε για τις ε, ε, κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Γαλλία ε, όταν έγινε η πρόταση για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Εμείς στην Ιρλανδία πρέπει να σας πω ότι πράγματι είδαμε τον κόσμο να στους δρόμους ακριβώς την ώρα που προτάθηκε αύξηση του ορίου ε, συνταξιοδότηση, του ορίου ηλικία για τη συνταξιοδότηση. Αυτό άρα δεν, δεν πρέπει να είναι χαρακτηριστικό μόνο τη Γαλλία, αλλά κάθε κράτο μέλου. Επίση, άλλα συστήματα, ε, μάλλον διαφορετικά συστήματα ή προϊόντα συνταξιδοτικά θα πρέπει να, να συζητηθούν, να μελετηθούν και ασφαλώς θα υπάρχουν και διαφορετικές λύσεις, αλλά θα ήθελα να δω και τι είδους απόψεις έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτά. Κύριο Κέστλερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ, συμφωνώντας με τους ε, προλαλήσαντες, να σημειώσω ότι όντως θεωρώ πως είναι δικής μας αρμοδιότητα στο ζήτημα της, ε, ε ξεοδοτικών συστημάτων. Θα πρέπει η δική μας δηλαδή Επιτροπή να αναλάβει την κατουσία ε, έκθεση. Αλλά τώρα επιτρέψτε να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που πιστεύω θα πρέπει να μας, θα μας απασχολήσουν. Θα υπάρξουν σημαντικέ αντιπαραθέσει απόψεων και όχι μόνο μέσα στην Επιτροπή μα, αλλά σε όλο το κοινοβούλιο και την ευρύτερη κοινωνία. Ένα ζήτημα θα είναι το πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι δικέ μα αρμοδιότητε. Αυτό θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα συζήτηση και την παράθεση με τους συναδέλφους και ίσως να μην τηρηθούν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο προκείμενο θέμα. Και όπως είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος νωρίτερα, θα πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα τα σχετικά με τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες με την ε, πολιτική για την απασχόληση παραδείγματι, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει αδήλωτη ή παράνομη λεγόμενη εργασία, μαύρη εργασία για την οποία δεν υπάρχουν ε, οι σχετικές εισφορές ή τα διαφορετικά συστήματα που επικρατούν ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. στη Γερμανία, Φερρυπίν, έχουμε ένα σύστημα συνταξιδοτικό το οποίο καλύπτει ο εργοδότης, αλλά υπάρχει και ζήτημα, ε, υπάρχουν μάλλον, υπάρχει και σύστημα που έχει να κάνει με τους δημόσιους υπαλλήλους όπου η ανταπόδοση ε, δεν είναι δεδομένη, δεν είναι ανταποδοτικό σύστημα. Επομένως, για μένα τίθεται το ερώτημα ως εξής. Εάν δεν φτάσω σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο, μπορώ να έχω μία ε, εντός αγωγικών συνταξιδοτική πρόνοια από την ιδιωτική μου ασφάλιση η οποία θα με καλύψει μέχρι ότου φτάσω στο όριο ηλικίας της σύνταξης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς απαραίτητα να έχουμε δεδομένη την απάντηση ή τον τρόπο με τον οποίο θα περάσει ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά όταν μιλούμε για ευελιξία, όταν μιλούμε για κινητικότητα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ε, ισχύσουν διαφορετικές λύσεις. Όλα αυτά νομίζω μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Και επίσης για μένα, και εδώ κλείνω, πολύ σημαντικό είναι στην ε, κατάσταση που μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος και την αναλογία μεταξύ ε, ενεργού πληθυσμού και συνταξιούχων, ίσως δεν είναι δεδομένο ότι η λύση θα βρίσκεται πάντοτε στην κρατική δημόσια σύνταξη, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μία ιδιωτική σύνταξη που θα συνοδεύει τον συνταξιούχο εν μέρη και θα μοιράζεται το βάρος, την, ε, την κάλυψη του συνταξιούχου με, μια δημόσια, με ένα δημόσιο σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο, να ενσωματώσουμε και στις εκθέσεις μας και περιμένω μια συζήτηση η οποία ήδη ε, προεξεγγέλλεται πολύ ενδιαφέρουσα. Η κυρία Κάστα έχει στη ζωή το λόγο, αλλά θα παρακαλήσω πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Nella traduzione ho dato un altro nome. Ε, ναι, άλλον μ' άκουσα. Τέλο πάντων να πω τρία πράγματα. Πρώτον, νομίζω ότι η συζήτηση που κάναμε καταδεικνύει ότι αυτή η ελιστική προσέγγιση θα πρέπει να διατηρηθεί και στα κοινωνικά θέματα και στα οικονομικά και στα θέματα της απασχόλησης. Οπότε η αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής της δικιάς μας θα πρέπει να υποστηριχθεί και να εξελιχθεί. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι το πράσινο βιβλίο είναι ένα κείμενο πλούσιο, ενδιαφέρον και συμφωνώ με αυτά που λένε διάφοροι συνάδελφοι ότι πραγματικά τα χρονοδιαγράμματα είναι λίγο κάπως ε, στενά ώστε να ζυμωθούμε έτσι μεταξύ μας στις σκέψεις και στις απόψεις. Και κάτι άλλο που νομίζω ότι είπαν και άλλοι συνάδελφοι Νομίζω δηλαδή ότι στις προκλήσεις που αναφέρουμε εμείς περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και το να κατανοήσουμε ότι το σύστημα που τώρα πια όλα τα συστήματα τα συνταξιδοτικά έχουν μια τάση να περάσουν από την κατανομή στην κεφαλαιοποίηση. Να ξέρουμε λοιπόν ότι σε περιόδους κρίσεως και τα δύο συστήματα παρέχουν ή προσφέρουν συστήματα επιβάρυνσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ανασφάλεια των νέων. Πολλές φορές μάλιστα έχουμε και το πρόβλημα της πρόσβασης στην συνταξιοδότηση. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας οπωσδήποτε το θέμα της γενιάς, της ηλικίας δηλαδή των εργαζομένων. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ευέλικτο να συνοδεύεται από συστήματα συνταξιδοτικά που λαμβάνουν υπόψη τους την ηλικία των εργαζομένων. Και για τις γυναίκες νομίζω ότι είναι κάπως ουδέτερη αυτή η πράσινη βίβλος σε σχέση με την απέτηση που ανέκυψε από τις ε, εργασίες μας για την αν όχι εναρμόνιση, τουλάχιστον προσαρμογή των συστημάτων γιατί αν δούμε τι ισχύει στις διάφορες χώρες μέλη θα δούμε ότι έχουμε πολλά συντοξιδοτικά συστήματα που συχνά οι γυναίκες λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις και πολύ συχνά όταν δεν τους αναγνωρίζονται δικαιώματα έχουν τις εισφορές χωρίς όμως αυτές τις φορές να φτάσουν στην ελάχιστη σύνταξη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε και μία εναρμόνιση όσον αφορά την σχέση μεταξύ ζωής και εργασίας. Και σε σχέση με αυτό που έλεγε και ο κ. Κοφεντεράτη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το, συγγνώμη που σας ε, ε, διακόπτω. Ε, σε εσάς λόγο μόνο για ελάχιστο χρονικό διάστημα, ένα λεπτό και συνεχίζεται πάπυρον. Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ δύο λόγια για τη συζήτηση αυτή, καταρχάς. Έχουμε το ζήτημα των προθεσμιών που ορίζει για την απάντηση του Κοινοβουλίου η Επιτροπή. Εάν θέλει με σοβαρότητα η Επιτροπή να συμμετάσχει στο Κοινοβούλιο στη διαβούλευση, 20 Νοεμβρίου δεν είναι καθόλου ρεαλιστική προθεσμία, γι' αυτό παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα να δώσετε μια παράταση σε αυτή την προθεσμία για τις διαβουλεύσεις. Διαφορετικά θα μπορέσει το Συμβούλιο να συμβάλλει στο διάλογο αυτόν, ίσως ούτε και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και, εν πάση περιπτώσει, για ένα τόσο περίπλοκο και σημαντικό θέμα δεν είναι δυνατόν να, να μην εκφέρει γνώμη το Κοινοβούλιο. Για τις αρμοδιότητες όλοι οι συνάδελφοι εδώ μίλησαν υπέρ της καθήλυνα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας για λόγους ουσίας, για λόγους ε, παρακολούθησης ε, των δομών που ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης. Όταν λοιπόν μιλούμε για better regulation αλλά και για καλή δουλειά, ασφαλώς θα πρέπει η έκθεση της κυρίας ε, Ομινρόιτεν να είναι εκείνη η οποία θα έχει την κατουσία να εξετάσει του θέματος. Και παρακαλώ και εσείς με, τους, με τις γνωριμίες σας στην Οικονομική, Κοινωνική, στην Οικονομική Επιτροπή, Οικονομική και Σωματική Επιτροπή, να πείστε τους συναδέλφους ότι η κατουσία καθήλυνα αρμοδιότητα ανήκει στη δική μας Επιτροπή. Για το περίπλοκο λοιπόν ζήτημα τώρα των όρων που επιλέγονται και μένω στο ερώτημα υπαριθμών 13 εάν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσδιορίσει συγκεκριμένες στατιστικές μια κοινή προσέγγιση για τις αυτόματες επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή και τις επενδυτικές δυνατότητες κτλ. Αυτό είναι ένα δείγμα μόνο πόσο περίπλοκη είναι αυτή η ερώτηση ή αυτές οι ερωτήσεις που θέτεται. Και θα ήθελα, αν είχαμε την ευκαιρία, να εμβαθύνουμε σε μια σειρά στοιχείων προκειμένου γιατί ναι, πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά πλήσεις μεταξύ των κρατών μελών σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την πραγματικότητα και τη στρατηγική που εισάγεται σε μια μεταρρύθμιση των συνταξιδοτικών συστημάτων, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δημογραφικές διαφορές. Επίσης, όταν έχουμε, έχουμε την πρόθεση έστω για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην υπόθεση αυτή, γιατί να μην μιλούμε για ένα ελάχιστο εισόδημα και ένα ελάχιστο όριο συντάξεων. Κοινού όρους ως προς το, ε, την έννοια του βαρέως επαγγέλματος, Φερρυπίν συστήματα για τον προσδιορισμό για, το, για κοινούς όρους ως προς το εξοδοτικό, ως προς τις συντάξεις ή επιπτώσεις ως προς το εισόδημα και όχι μόνο αξιολόγηση των, των δημοσιονομικών ως ε, προϋπόθεση για την ε, βιωσιμότητα ενός εξωτικού συστήματος, αλλά και όλους τους άλλους οικονομικούς παράγοντες, όλες τις άλλες οικονομικές παραμέτρους και επίσης θα συμφωνήσω και εγώ με τη συνάδελφα που μίλησε νωρίτερα για την ανισότητα, την απουσία ισότητας μεταξύ των φύλων στην υπόθεση της απασχόλησης και της σύνταξης, πράγμα το οποίο ε, αγνοεί η πράσινη βίβλος, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί. Έτσι λοιπόν, όταν ε, ξεκινάμε μια οριζόντια διαβούλευση για το θέμα αυτό, δεν θα ήταν σκόπιμο και η κινητικότητα της αποταμίευσης ε, να συζητηθεί εν ώψη συστημάτων ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων και με μια καλή ανταπόδοση. Η απόδοση καλύτερα. Δεν έχουμε λοιπόν επαρκή χρόνο και ξέρω πολύ καλά ότι ε, ε, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση οι προσκεκλημένοι μας ε, όταν τους ζητήσω μέσα σε δύο λεπτά να μας απαντήσουν σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας πιέζει και ενδεχομένως όταν έρθει η ώρα για τη συζήτηση επί της ουσίας της εκθέσεως της κυρίας Ομενρόιτεν να τους δώσουμε πάλι την ευκαιρία να τους καλέσουμε και πάλι να μας μιλήσουν. Κύριε Φίσερ, πρώτα απ' όλα, κύριο ερώτημα κέριο ερώτημα, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια παράταση τη προθεσμία για το Κοινοβούλιο. Γιατί δεν είναι δυνατόν το Κοινοβούλιο σοβαρά να συζητήσει το θέμα αυτό με την προθεσμία που έχει το ορίσει. Μόνο σε ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ, γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να δώσω άμεση απάντηση στην ερώτησή σας. Δεν είναι δική μου η απόφαση. Πρέπει να σας πω ότι ε, οι τέσσερις α, ε, μήνες είναι μία περίοδος όντως πιο σύντομη από την περίοδο που προβλέπεται συνήθως κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Καταγράφω πάντως το αίτημά σας και θα σας δοθεί σύντομα μία απάντηση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η συζήτηση που έγινε εδώ ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αναφερθήκατε σε πολλά και σημαντικά ζητήματα. Δεν λέω ότι καλύπτονται όλα τα ζητήματα στην Πράσινη Βίβλο, πάντως καταγράφω τα όσα είπατε, το ζήτημα τη αβεβαιότητα, το ζήτημα της Μαύρη μαύρης οικονομίας, της εργασία, εργασίας, το ζήτημα της οικογενειακής πολιτικής, ισότητα των φύλων, το ζήτημα της περίθαλψης. Τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ σχετικά με τη διαμόρφωση των μελλοντικών συνταξιωτικών συστημάτων. Επίσης καταγράφω τα όσα είπατε για την ε, αρμοδιότητα και για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται αυτή τη στιγμή να επιφέρει μια προστιθέμενη αξία. Δεν θέλουμε εμεί απλώς όντως να φέρουμε το ζήτημα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πέρα από αυτό. Θέλουμε όντως αυτό να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τους πολίτες και να βοηθήσει αστικά τις κυβερνήσεις να διαμορφώσουν καλύτερα τα συνδοξικά του συστήματα. Στα δύο λεπτά απλώς που είχα στη διάθεσή μου, ολοκληρώνοντα λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίε της δική μου τη μονάδα είναι στη δική σα τη διάθεση προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε και εσάς να διαμορφώσετε μια άποψη στα πλαίσια τη συζήτηση αυτή. Πάντως μετά από την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων που έγινε προσβλέπω σε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, μια συζήτηση που με σίγουρο θα είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για του τέσσερι μήνε τη διαβούλευση, όμω μην ξεχνάτε ότι ένα μήνα ήταν μέσα στο καλοκαίρι, ήταν μήνα διακοπών. Και στην επόμενη συνεδρίασή μα, στην επόμενη συνεδρίαση Επιτροπή, ο επίτροπο θα έρθει εδώ, επομένω θα του απευθύνουμε άμεσα την ερώτηση αυτή, το αίτημά μας. Ο κύριος Whitehouse τώρα έχει τον λόγο. Δύο λεπτά επίσης. Δεν είναι δικός μου ρόλος να τοποθετηθώ για την εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκ μέρους του ΟΣΑ απλώς θα ήθελα να πω ότι ε, αξιολογούμε τι χώρες του ΟΣΑ στην συνταξιωτική της πολιτική και μία μελέτη θα δημοσιευθεί το Δεκέμβριο η οποία θα αναφέρεται ακριβώς και στο ζήτημα αυτό της ηλικία συνταξιοδότησης, στο ζήτημα των ε, εξελίξεων στο προσδόκιμο ζωής, ε, στις ε, καινούργιες προβλέψεις που μπορεί να υπάρχουν βάσει του προσδοκίμου ζωής και θα αναφερόμαστε επίσης στο γεγονός ότι ε, υπάρχουν διάφορα κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, η Ιταλία που μεταρρυθμίζουν το στεξιωτικό σύστημα το προκειμένου να εναρμονίζεται απόλυτα με τις εξελίξεις και τις προβλέψεις στο προσδόκιμο ζωής. Επίσης θα έχουμε ένα ξεχωριστό έγγραφο όσον αφορά τις γυναίκες και τα συνταξιωτικά συστήματα και στα πλαίσια του εγγράφου αυτού θα ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα των φύλων και ιδίω με την ε, μεταχείριση εκείνων των γυναικών οι οποίες κατά τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους είχαν συγκεκριμένε ε, περιόδους ε, κατά τις οποίες δεν εργάζονταν, βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας. Θέλουμε κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τι ε, χώρε και τι κυβερνήσει να διαμορφώσουν στα εξωτικά συστήματα τα οποία θα τα περισσότερο στο διαφορετικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι άνδρε και οι γυναίκε στι κοινωνίε. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Όντω πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Όμεν Ρόιτεν, έχετε το λόγο, ναι, τον έχετε, αλλά να είστε πάρα πολύ σύντομοι, παρακαλώ. Θα είμαι όντως σύντομη, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που παρατήρησα κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι ότι πολλοί από αυτούς πήραν το λόγο. Αναφέρθηκαν σε διάφορα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την προοπτική της δικής τους χώρας, με μια εθνική στρατηγική βασικά. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν και κάποιες συζητήσεις με συγκεκριμένα άτομα στην Επιτροπή αυτή, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια αξιοπρεπή έκθεση, η οποία θα έχει μια κοινή θέση θα έχει μια κοινή κατεύθυνση. Όσον αφορά το ζήτημα τώρα των φύλων, αυτό το οποίο πρέπει να επιτύχουμε είναι να εξασφαλίσουμε μια υποστήριξη της γυναίκες παντού στην Ευρώπη. Πρέπει η προστιθέμενη αυτή η κοινοτική αξία να ωφελεί και τις γυναίκες. Έχουμε δει επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένε αποφάσεις υπέρ των γυναικών, αποφάσεις που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κάτι ακόμα. Όσοι έχουν το καθεστώ τη απασχό... μερικής και αυτοί θα πρέπει να χαίρουν μια καλύτερη μεταχείρισης στο μέλλον. Στη δική μου χώρα έχουν ήδη επιτευχθεί κάποια πράγματα δεν λέω ότι δεν έχει συμβεί αυτό και από άλλε χώρε, δεν λέω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδο γενικότερα. Πάντω, εκκρεμούν ακόμα πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν όσον αφορά δηλαδή και τη μερική απασχόληση. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή την πράσινη βίβλο και να προσπαθήσουμε απλώ χρησιμοποιώντα αυτή τη βίβλο να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε κενά τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στην δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρέπει απλώ να δούμε τι πρέπει να γίνει πού εντοπίζεται η προστιθέμενη αξία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού πρέπει τα κράτη-μέλη με τη σειρά τους να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να διορθώσουν την κατάσταση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον και με την ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να κάνουμε μια καλύτερη οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων Ξέρω ότι δεν σας έδωσα πάρα πολύ χρόνο για να εκφραστείτε. Ελπίζω όμως ότι καταφέρατε να ακούσετε και τους περισσότερους συναδέλφους σε αυτή την Επιτροπή. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο υπαρεθμόν 10, με θέμα την βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστεί η πρόεδρος του Δερμηνής που θα δουλέψουν 10 λεπτά παραπάνω. Το λόγο έχει ο κύριος Κάζα, ο οποίος θα υποβάλει μια γνωμοδότηση ε, για την έκθεση την οποία θα καταθέσει ο κύριος Φέιο για την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που είναι η αρμόδια επί τη ουσία. Κύριε Κάζα, έχετε το λόγο. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι όσο σύντομο γίνεται. Όπως ξέρετε, η έκθεση της ΕΙΚΟΝ αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Έχουμε 8 συστάσεις. Η γνωμοδότηση αποβλέπει στην περαιτέρω ενδυνάμωση αυτών των συστάσεων περιλαμβάνοντα την προοπτική της απασχόλησης. Μίλησα με διάφορους συναδέλφους στην Επιτροπή μαζί με τους Κιώδη. και θα έπρεπε να είμαστε πολύ σύντομοι λόγω του περισμού του 1500 χαρακτήρων. Παρ' όλα αυτά ε, θα μπορούσαμε να επεκταθούμε στα θέματα αυτά μέσω τροπολογιών. Πρώτον, λοιπόν τα εξή. Καταρχήν τη θέσπιση ενός πλαισίου παρακολούθησης ή εποπτεία που θα, αφορά δύο πυλώνες, οικονομικές και οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Θα θέλουμε επίσης να ενισχυθεί και ο ρόλος της Επιτροπής απασχόληση ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της διασυνοριακής εργασίας. Θα θέλαμε βεβαίω να συμμετάσχει όσο περισσότερο γίνεται το κοινοβόλιο στην εποπτεία αυτών των πολιτικών και τέλος η έκθεση ΕΚΟΝ προβλέπει κάποιες ποινές σε περίπτωση που δεν υπάρχει τήρηση κάποιων κανόνων σε σχέση με τα θεωρητικά ταμεία κτλ. Θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό γιατί τα θεωρητικά ταμεία σε σχέση, σε σύνδεση με την ε, απασχόληση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ. Θεωρούμε ότι το σύστημα των κυρώσεων και των ποινών θα πρέπει ξεκάθαρα να διακρίνει μεταξύ κονδυλίων που καταγράφονται στα εθνικά στου εθνικού προπολογισμού και τα κονδύλια τα οποία αφορούν του μεμονωμένου πολίτε και εργαζόμενου. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η, ιδέα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να απορριφθεί. Οπότε, καταλήγοντας να πω ότι προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτή την γνωμοδότηση και βεβαίως αναμένω με χαρά τις ε, τροπολογίες που θα καταθούν και που θα συζητήσουμε ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, ε, ο κύριος Σαρκάς και μετά ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης από τους σοσιαλιστές είναι η κυρία Ράτχη. Η κυρία Ράπτη, η οποία είναι στην Ελλάδα. Όμως μου έδωσε ένα έγγραφο το οποίο θα σχολιάσω. Καταρχήν μου είπε ότι λυπάται που απουσιάζει και θα πρέπει και εμείς βεβαίως να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες που θα πρέπει να τονίζουν τα εξής. Τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών σχεδίων ε, σύγκλησης και της στρατηγικής 2020 την συμπλήρωση των ε, προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στόχους για την απασχόληση θα πρέπει να τονίσουμε και τη σημασία του έψω σχέση με το ΕΚΟΦΗΝ. Θα πρέπει να υπάρχει ο στόχος της κοινωνικής πολιτικής μέσω αυτών των πυλώνων που αναφέραμε προηγουμένως και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την εργοποίηση της κοινωνικής ρήτρα ή δικλήρας που περιλαμβάνει η συνθήκη της Λισαβόνας ώστε να έχουμε πράγματι ουσιώδεις ε, εγγύηση ώστε να περιλάβει στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον πυρήνα των πολιτικών της, το θέμα τη εργασία και της απασχόλησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ο κ. Κοφεράτη και μετά κυρία Γκρούνη. Σύντομα, Πρόεδρε. Το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι θετικές και καθορίζουν τα σημεία προτεραιότητας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αναπτυχθούν. Βεβαίω υπάρχει στη συνέχεια το θέμα της συντακτικής διάταξης ή διάσταξης διά... μεγέθους τόσο πάνω του κειμένου. Υπάρχουν και άλλα σημεία που θα πρέπει να αναφέρουμε νομίζω και προσωπικά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο αλλά νομίζω θα το αναφέρουμε και αυτό στην ε, συζήτηση με τις τροπολογίες, θα πρέπει να δώσουμε κυρίως έμφαση σε αυτές τις δύο πτυχές που ανέφερε και προαλήσαντας, επειδή η τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και κυρίως η χρήση του Συμφώνου Σταθερότητας ως στοιχείου που οθεί στις επενδύσεις και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε δηλαδή θα πρέπει να το θεωρήσουμε όχι ως μόνο μια μεταβατική λύση αλλά προς ένα σταθερό σημείο της οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης άλλο ένα σημείο το οποίο είναι επίμαχο όσον αφορά τις συζητήσεις για την κατανομή του εισοδήματος, δηλαδή για την ποιότητα στην ουσία του εισοδήματος που συνδέεται με τις επιδόσεις και με τους μακροπρόθεσμους στόχους να πω ότι αν δεν λύσουμε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που είχαν παλαιότερα στην Ευρώπη και που μεταξύ άλλων πριν από 20 χρόνια είχε οδηγήσει τον Ζακ Τελόρ να εκδώσει την Λευκή Βίβλο για επενδύσεις μικρομεσαίες σε μεσαίο και μακρόχρονικό διάστημα όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στα βραχυπρόθεσμα κέρδη ξέχασαν την αρχική τους αποστολή σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο του Ζακ Τελόρ. Οπότε θεωρώ ότι αυτό, δηλαδή το να επικεντρωθούμε σε αυτά τα στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ένα άλλο καινοτόμο στοιχείο τη οικονομική διακυβέρνηση. Κύριε Γκρούνη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω να συγχαρώ τον κύριο Κάσα για το σχέδιο γνωμοδότης το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ συνετό. Θα ήθελα μόνο να επιμείνω στο σημείο 7 γιατί είναι αλήθεια το να επιβάλλουμε κυρώσεις μέσω των ιδρυτικών ταμείων αυτό είναι νομίζω καταρχήν κατά προσδόκητο και σε τελική ανάλυση θα αποτρέψει κάποιους Ευρωπαίους από το να επωφεληθούν από κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζονται απαραίτητα. Αναφέρει και την ε, φοροδιαφυγή και την απάτη, τη φορολογική απάτη, όπως επίσης και την κοινωνική απάτη στην γνωμοδότησή του. Η κοινωνική απάτη θα πρέπει να τονιστεί επειδή νομίζω σε τελική ανάλυση αποτρέπει τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια να αποφεληθούν από όλα αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το σημείο 3 να πω ότι μιλάμε για συστήματα πρόνοιας και σύνταξης όπου θα πρέπει να προσθέσουμε και την κοινωνική πρόνοια εδώ ως όρο. Αυτά πρόεδρε ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα έχουμε βεβαίω την ευκαιρία να δούμε τι τροπολογίε και να δούμε πιο συγκεκριμένα τα σημεία αυτά. Εγώ απλά και μόνο θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Α, κυρία Μάρκη, με συγχωρείτε, σα ξέχασα. Πώς μπορέσατε. Ναι, μπόρεσα. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη κι εγώ. Η απάντησή μας στην οικονομική κρίση νομίζω δεν θα πρέπει να στηρίζεται υπερβολικά στις μεταρρυθμίσεις και στις κυρώσεις. Συμφωνώ με τον συντάκτη της νομοδότησης ότι εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μεταρρυθμίσεις των συστημάτων ε, πρόνοιας, ε, σταξιδότησης κτλ. Είναι καλή που το κείμενο και συμφωνώ με την, άποψη, με την άποψή σας για το σύστημα των κυρώσεων και είμαι καθόλου βέβαια ότι το σύστημα κυρώσεων θα είναι χρήσιμο. Σε τελική ανάλυση θα ζημιωθούν οι πολίτες. Θα ζημιωθούν δηλαδή αυτοί που θα χάσουν τη δουλειά τους και θα πρέπει να φύγουν σε άλλες χώρες. Και τελικά νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος αυτή. Αυτά πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, επανέρχομαι στο σημείο που θα ήθελα να πω από την αρχή. Δηλαδή το καθεστώς κυρώσεων το ανέφεραν και το σχολήσαν διάφοροι συνάδελφοι. Θα πρέπει ενδεχομένω να δούμε τη διατύπωση, γιατί εδώ έχουμε την εντύπωση ότι η μόνη κύρωση που δεν θέλουμε είναι αυτή που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν είναι αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά νομίζω η σύνταξη αυτό αφήνει να Νομίζω λοιπόν ότι το ενδεχόμενο αφαίρεσης δικαίωμα ψήφου για κάποια σημαντική χρονική περίοδο νομίζω αντιβαίνει στην ίδια την της αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η δημοκρατία. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα πεδίου εφαρμογής των κυρώσεων αλλά συμφωνώ με αυτό που λέγατε προηγουμένως ότι μέσω αυτών των κυρώσεων θα επιτρέψουμε και άλλες κυρώσεις. Τώρα, επειδή συγκεκριμένα έχουμε να κάνουμε με ένα μια έκθεση που αφορά τα εργαλεία της διακυβέρνηση, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι κοινό μεταξύ ΕΦΣΚΟ και ΕΚΟΦΗΝ. Δηλαδή ε, το Συμβούλιο και το ΕΚΟΦΗΝ να συνεργαστούν από κοινού. Κάποιες άλλες παρατήσεις να κάνω επίσης. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και τον κίνδυνο της δημοσιονομικής σταθεροποίησης η οποία θα μπορούσε να γίνει εις βάρος της κοινωνικής συνοχής όπως είδαμε ας πούμε στην Ελλάδα. όπου αποφάσισαν τη μείωση κατά 15% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και υπάρχει μια κοινωνική ισορροπία η οποία κατά την άποψή μου είναι ένα διακυβόμενο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος. Τώρα για τη στρατηγική των μακροχρόνιων επενδύσεων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στα πλαίσια μιας διακυβέρνησης ε, σύμφωνης με το 2020 και τη στρατηγική νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν νομίζω είχε πει ότι δεν αρκεί να έχουμε ένα άρθρο 9 για να αποτιμήσουμε τις, επιπτύ, τις επιπτώσεις. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτά που κάνουμε δημιουργούν απασχόληση, δημιουργούν θέσεις εργασίας και επανεχόμενοι σε αυτά που είπε ο κ. Κομφεράτη Κατά τη διάρκεια τη οικονομική και Νομισματικής Ένωσης ε, θα έπρεπε, είπε ο κ. Κοφεράτη, να έχουμε καθορίσει κάποιους στόχους που αφορούν βεβαίως τα οικονομικά αλλά και κάποιους στόχους που αφορούν την ε, απασχόληση δηλαδή που προβλέπουν συγκεκριμένα επίπεδα απασχόληση των νέων, επίπεδο ανεργίας κλπ. κλπ. Στόχοι δηλαδή και στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της, της καλής, της χρηστής οικονομικής κοινή διακυβέρνησης. Μετά έχουμε και το θέμα της, της ανταγωνιστικότητας των χωρών μελών επειδή δεν θα θέλαμε να εξασθενήσει το κοινωνικό μοντέλο κάποιας χώρας και αν υπάρχει μεγάλη απόκληση ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων οικονομιών, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε μπορούν να αναπτύξουν το κοινωνικό του μοντέλο και άλλε χώρε οι οποίε δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε νομίζω θα πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ από τη σκοπιά αυτή την γνωμοθέτησή σας αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε περαιτέρω. Αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και θα τα έχουμε καταφέρει μια χαρά με τον χρόνο και εσύ θα έχετε το λόγο. Ναι, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, Πρόεδρε. Νομίζω ότι άκουσα του συναδέλφου, κατέγραψα τι προτάσει και θα τι συνδυάσω με τι δικέ μου τροπολογίε. Αν δεν κάνω λάθο, ήδη είχα 7 τροπολογίε Αύριο το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε μια επισκόπηση όλων αυτών των ιδεών αύριο όταν θα εκπνεύσει η προθεσμία για τις τροπολογίε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, συμβολή σας επειδή ακολουθήσαμε τέλεια τον χρόνο. Η νύχτα βοηθάει. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ.